Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Με την τακτική συνάντηση της Επιτροπής ΙΝΤΑ όλοι θα λάβατε το σχέδιο μέτρησης διάταξης. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε σχόλια από αυτής. Όχι. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν η μέτρηση διάταξη. Το σημείο 2. Τώρα ανακοινώσει του Πρόεδρου. Σύντομο θα είμαι. Ο συνήθω τη συνεδρίαση είναι online. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ όσου βρίσκονται και μας παρακολουθούν μάλλον διαδικτυακά από το Ταλίνινο στη Θεσσαλονίκη και τη Λισαβόνα. Υπάρχει διερμηνία, οπότε παρακαλώ να είστε σαφείς στις παρεμβάσεις και όχι υπερβολικά γρήγοροι και ευθύ αμέσω θα περάσει στο σημείο 3 τη ημερήσια διάταξη. Οι εμπορικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Αυστραλία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκονται εδώ μαζί μα κάποια μέλη του Κοινοβουλίου τη Αυστραλία. Ο Κέβιν Έντριου είναι εδώ μαζί μα, επικεφαλή αντιπροσωπεία αυτέ. Ήταν υπουργό ε, σε διαδοχικέ κυβερνήσει, κυρίω ε, υπουργό άμυνα αλλά και βέβαια ε, μέλος του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου για πολλά χρόνια. Καλώς ήρθατε. Βεβαίω η Αυστραλία και η Ευρώπη έχουν στενές σχέσεις αργήσαμε ε, να ξεκινήσουμε συζητήσεις εμπορικές με την Αυστραλία διότι έχουμε ήδη μια πολύ στενή σχέση Έχουμε κοινωνίες ε, ε, που είναι, έχουν αρκετά κοινά σημεία, παρότι βεβαίως βρισκόμαστε πολύ μακριά γεωγραφικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή ΙΝΤΑ τον Νοέμβριο του 2017 επισκέφθηκε το Σίδνεϊ και την Καμπέρα. Αμέσως ε, μετά την έγκριση ενός ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η Αυστραλία επίσης έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις στο πολυμερές σύστημα. Ένα πολυμερές σύστημα το οποίο, όπως ξέρετε, ε, απειλείται αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε κάποιες, κάποιους νέους δασμούς που θα επιβληθούν από τις ΗΠΑ, παραδείγματος χάρη τις επόμενες μέρες και αυτό θα οδηγήσει σε κλιμάκωση και νέες απειλές για το πολυμερές αυτό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθεροποιήσουμε ένα εμπορικό σύστημα που να βασίζεται σε κανόνες και η εμπορική συμφωνία με την Αυστραλία συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Ο εισηγητής μας για το σύστημα αυτό είναι ο Ντανιέλ Κασπάρη. Θα του δώσω τον λόγο ευθύ αμέσω. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι φίλοι από το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω τη δική σας γλώσσα, ε, αλλά εάν δεν καταλαβαίνετε τα αγγλικά μου υπάρχει διερμηνία προς τα αγγλικά. Το Μάιο πέρσι το Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει τι πραγματεύσει για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυστραλία. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο πέρυσι. Είμαστε ακόμα λοιπόν στην αρχή, αφενός. Αφετέρου, έχω την εντύπωση ότι και οι δύο πλευρές έχουν, επιδεικνύουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα, να έχουμε καλές διαπραγματεύσεις. Έτσι λοιπόν το έτος που πέρασε ήταν εξαιρετικά παραγωγικό προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς έχουμε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας ε, στην, ε, στο πλαίσιο σύμπραξης με την Αυστραλία το 2018 είναι ε, ο 18ος εταίρος, εμπορικός εταίρος σε αγαθά και εμείς είμαστε ο δεύτερος εταίρος μετά την Κίνα για την Αυστραλία. Είχαμε τέσσερις γύρους διαπραγματεύσεων, τελευταίο εκ των οποίων τον Ιούλιο φέτος και ο επόμενος γύρος προβλέπεται 14 με 18 Απριλίου στην Καμπέρα και στη συνέχεια το Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες. Ε, η ιδέα αυτή τη εμπορική συμφωνία είναι να διευκολύνει το εμπόριο για τα βιομηχανικά προϊόντα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυστραλία, μειώνοντα ε, τα τεχνικά εμπόδια και βελτιώνοντα τι υπηρεσίε και τι επενδύσει. Ε, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια εμπορικά εμπόδια που πρέπει να προσπαθήσουμε να απαλείψουμε. τα, τα δασμοί ε, παραδείγματο χάρη στον τομέα των αγαθών, το θέμα των δημοσίων προμηθείων. Υπάρχουν μια σειρά αποστήματα, τα χημικά, μεταποιημένα προϊόντα, υπηρεσίε, ε, όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Θέλουμε να προστατεύσουμε και ευάλωτου τομεί όπω η γεωργία, μεγιστοποιώντα ε, τα, τα ωφέλη από το άνοιγμα τη αγορά, χωρί όμω να πλήττονται ευαίσθητα προϊόντα. Δεν θέλουμε λοιπόν να πλήρη απελευθέρωση των ε, ε, εμπορική απελευθέρωση των γεωργικών προϊόντων, διότι ορισμένε φορέ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει. Θέλουμε επίση οι γεωγραφικέ ενδείξει να προχωρήσουν. Είναι ένα ζήτημα που οι εμπορικοί μα εταίροι δεν ε, του αρέσει ιδιαίτερα, αλλά ορισμένε φορέ ε, η καινοτομία εισάγεται από το εξωτερικό. Ε, θα ήθελα να ξέρω επίσης ε, ποιες είναι δικές σας απόψεις, οι απόψεις της για το Πώ βλέπετε αυτέ τι εμπορικέ σχέσει, πώ βλέπετε την υποστήριξη που υπάρχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση στο Κοινοβούλιο τη Αυστραλία. Έχετε μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα αυτή τη στιγμή και η Κίνα παρουσιάζει ενδιαφέρον για μας βέβαια. Εσεί έχετε ήδη ε, έτσι, αποκομίσει κάποια πρώτα διδάγματα. Όταν βλέπουμε τι επενδύσει των Κινέζων στην Αυστραλία με βάση το νέο FDA, εμεί αντιμετωπίζουμε το ζήτημα των επενδύσεων της Κίνα. Ε, που είναι καλοδεχούμενε ε, στην Ευρώπη, απ' την άλλη υπάρχουν ανησυχίε ε, σε κάποιου συγκεκριμένου κλάδους και για κάποιε συγκεκριμένε επιχειρήσει. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ε, πέρα από τι διμερεί εμπορικέ σα επαφέ πώ βλέπετε εσεί τη σχέση μα με την Κίνα και πώ μπορεί η Αυστραλία να είναι μια γέφυρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση προ την περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Αναμένω την παρέμβασή με πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον Κέβιν Άντριους. Και στη συνέχεια δώσει το λόγο στην Ιωάννα Βάιν. Παρακαλώ. Um, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου και προνόμιο να βρίσκομαι εδώ με την αντιπροσωπεία μου. Χθε είχαμε σημαντικές συναντήσεις με πολλές επιτροπές και μέλη του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συνεχίσω με ελπίζω τις θερμές σχέσεις μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ε, μαζί μας είναι και ο πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Προσβλέπουμε σε αυτές τις συνεχιζόμενες συζητήσεις όπως σας είπα. Η Αυστραλία είναι έθνος που πάντοτε ασχολείται με το εμπόριο και για 200 χρόνια η ευημερία μας στηρίχθηκε στην ικανότητά μας του συναλλάσσεις εμπορικά με άλλες χώρες στον κόσμο. Επίσης ε, είμαστε ένα έθνος το οποίο δεσμεύεται σε διεθνείς κανόνες. Η ευημερία όλων των λαών ε, προχωρά μέσα από τη συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες. Τρίτον, είμαστε μια χώρα που έχει κοινές αξίες με την Ευρώπη τις συμμεριζόμεθα γιατί το υπόβαθρό μας είναι ευρωπαϊκό αφού οι περισσότεροι Αυστραλοί ακόμα και σήμερα ε, μετανάστευσαν από την Ευρώπη και στη δική μου εκλογική περιφέρεια υπάρχουν πολλοί Έλληνες, Ιταλοί, Ολλανδοί και από ε, των πολίτες των πρώην ε, ανατολικών, χωρών του Ανατολικού Μπλοκ. Έτσι λοιπόν έχουμε κοινού δεσμούς και θα συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον, όπως είπε ο διακεκριμένος ομιλητής, η Ευρώπη είναι ο δεύτερος σε μέγεθος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας. Και παρόλο που γίνονται συζητήσεις που είμαστε παρατηρητές, εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο όγκο συναλλαγών. Αυτό είναι σημαντική σχέση που θέλουμε να την βελτιώσουμε και στο μέλλον. Ανεξάρτητα από τους συναισθηματικούς δεσμούς που μπορεί να έχουμε προς κάποιο έθνος, είμαστε και ορθολογιστές, πρακτικοί άνθρωποι, προσανατολισμένοι στο μέλλον, όχι στο παρελθόν. Το μέλλον συνεπάγεται πολύ στενές και αυξανόμενα θερμές σχέσεις με την Ευρώπη και σε ό,τι αφορά τις πολιτισμικές αξίες και τις αξίες μας σε έναν κόσμο αβέβαιο αλλά και σε σχέση με τα πρακτικά στοιχεία του εμπορίου. Το λέω αυτό εισαγωγικά γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι προερχόμεθα από παρόμοιες αφετηρίες σε ό,τι αφορά τις αξίες που φέρνουμε στο εμπόριο και τις διαπραγματεύσεις και πιστεύουμε σε ένα σωστό ρυθμιστικό σύστημα που δεν το συμμερίζεται αναγκαστικά και, και κάθε άλλο κράτος στον κόσμο. Εμείς όμως θεωρούμε ότι αυτό είναι μια κοινή αξία Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντιπροσώπων της, τους. Έτσι λοιπόν θέλουμε εμπορικές συμφωνίες, ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν ε, σωστά οι συζητήσεις. Είχαμε τέσσερις γύρους, ο πέμπτος θα γίνει τον Οκτώβριο στην Αυστραλία και πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, μια συνολική εμπορική συμφωνία που θα είναι αμοιβαίο όφελος. Υπάρχουν ε, βεβαίως ε, ευαίσθητα θέματα. Η γεωργία είναι ένα τέτοιο σημαντικό θέμα και ως γιος γεωργού, που παντρεμένος με κόρη γεωργού, καταλαβαίνω τι, ε, τι θέλουν οι γεωργοί. Είτε είναι στη Βέλγιο ή στην Πολωνία ή οπουδήποτε στην Ευρώπη ή στο Κουίνσλαντ ή στη Βικτόρια, ε, στις πολιτείες της Αυστραλίας. Όλοι ενδιαφέρονται στο στα προϊόντα τους, στη, στο μέλλον, στη, στο δίκαιο εμπόριο. Εμείς μπορέσαμε να επεξεργαστούμε τις δυσκολίες με άλλες χώρες του κόσμου, την Κίνα που αναφέρθηκε με την οποία έχουμε συμφωνία, με την Ιαπωνία έχουμε συμφωνία και άλλες χώρες στον κόσμο. Μπορούμε να τις επεξεργαστούμε αυτές τις δυσκολίες γιατί ε, σεβόμαστε ε, την, ε, το υπόβαθρο και την ιστορία κάθε χώρας και μπορούμε να βρούμε πάντοτε, να βρίσκουμε συμβιβαστικές λύσεις που θα ωφελούν όλους. Και αυτό ισχύει και για την Ευρώπη και για την Αυστραλία και για τους λαούς που εκπροσωπούμε. Ερχόμαστε με καλή θέληση, με γνήσια επιθυμία να συνάψουμε μια νέα συμφωνία αφού πιστεύουμε ότι μέσα από το εμπόριο και την, καθ' όλη την ιστορία μας των 200 ετών η Ευρώπη έπαιξε μεγάλο ρόλο και μέσα από το εμπόριο η ευημερία ε, της χώρας μας αναβαθμίστηκε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την Κίνα, ε, όπως με παρακαλέσατε. Η Κίνα προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες και μεγάλες προκλήσεις. Για κάποιο διάστημα, νομίζω ότι εμείς στη Δύση ιδιαίτερα θεωρούσαμε ότι καθώς ε, ε, ενισχύεται οικονομικά η Κίνα θα γινόταν και πιο φιλελεύθερη. Αυτό είναι μια υπόθεση που δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει πλέον. Έχει διαφορετικό καθεστώς, εμείς έχουμε εμπορικέ σχέσεις με την Κίνα, θέλουμε να συνεχίσουμε, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό με τα μάτια ανοιχτά και γνωρίζομαι ε, τα γεγονότα που συμβαίνουν σε σχέση με την Κίνα. Υπάρχει τώρα εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνα και ΙΠΑ ε, που ελπίζομαι να ε, σταματήσει σύντομα γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Βλέπουμε ότι επηρεάζεται και ο κλάδος της, το, της παραγωγής ε, και έχει και δευτερογενείς επιπτώσεις ε, που αφορούν τους πόρους. Ε, Εμεί θέλουμε να φροντίσουμε οι επενδύσεις να μην αντίκυνται στα εθνικά μας συμφέροντα. Έχουμε επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες. Στην Αυστραλία γνωρίζομαι ότι φροντίζομαι να μην υπάρχει στρέβλωση του εμπορίου με την κάθετη, για παράδειγμα, ολοκλήρωση ε, ε, και τη διασύνδεση παραγωγής ε, και εμπορικών αλυσίδων. Αν, για παράδειγμα, μια εταιρεία αγοράσει όλα τα επίπεδα αυτής της κάθετης ολοκλήρωσης, τότε δημιουργείται στρέβλωση χωρίς να μπορεί να παρεμβαίνει ο παραγωγός. Παρακολουθούμε λοιπόν πάρα πολύ τι συμβαίνει ως προς αυτό. Επίσης, θέλουμε να φροντίσουμε, να εξισορροπήσουμε τις στρατηγικές μας ε, ε, πολιτικές. Ε, ε, μας ε, ενδιαφέρει, για παράδειγμα, η μας ενδιαφέρει στην ε, διαδικασία του 5G ε, να προσεγγίσουμε περισσότερα την Ευρώπη ε, που, με την οποία έχουμε πολύ πιο κοινά στοιχεία από ότι με την Κίνα η οποία είναι ε, εταίρος μας, αλλά θέλουμε, ιδιαίτερα σε σχέση με την Κίνα, να αντισταθμίζουμε και τα στρατηγικά μας συμφέροντα, τα οποία είναι πραγματικά και έτσι έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και επαγρυπνούμε ε, ως προς αυτό, παράλληλα με τις προσπάθειες για μεγαλύτερη ευημερία στο μέλλον όλοι θα ωφεληθούν βεβαίως ε, αν υπάρξει μια διεθνώς συμφωνηθήσα ε, ρύθμιση ε, θεμάτων εμπορίου. Αυτό θα ωφελήσει όχι μόνο την Αυστραλία και την Ευρώπη αλλά και την Κίνα. Και ε, ελπίζω να πιστεί η Κίνα ότι είναι προς το συμφέρον της, ότι να υπάρχει ένα τέτοιο διεθνές σύστημα κανόνων για το εμπόριο κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ, όπως είπα και στην αρχή. Νομίζω ότι αυτό είναι, συμβάλλει στην ε, θερμή και ε, συζήτηση που αρχίσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των καλών μας σχέσεων και ελπίζω να προχωρούμε όλο και καλύτερα και για την Ευρώπη και για την Αυστραλία στο μέλλον. Ε, αν κάποιοι συνάδελφοι επιθυμούν, δικοί μου επιθυμούν να παρέμβουν, παρακαλώ. όλοι λένε όχι. Ευχαριστούμε πολύ τον Κέβιν Άντριους. Και τώρα ο λόγος του συναδέλφου δύο λεπτά ο καθένας. Η Μακουλάδα πρώτη από την Ισπανία. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, μου άρεσε πάρα πολύ η παρέμβασή σας. Όντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία ε, μοιράζονται ε, μια κοινή θεώρηση ό,τι αφορά το διεθνές, ε, τη διεθνή πολυμερή τάξη πραγμάτων. Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα σχετικά με αυτό το πολυμερή χαρακτήρα. Ε, πώς βλέπετε σε αυτή τη στιγμή την κατάσταση, την περίπλοκη κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε σε σχέση με τον ΠΟΕ και πώς βλέπετε ε, εσείς να μπορούμε να φτάσουμε σε μια πολυμερή συμφωνία και μια μεταρρύθμιση και πώς ενδεχομένως η Κίνα θα εμπλακεί σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείτε στην Αυστραλία ε, τι δυνατότητες έχει το Κοινοβούλιο ε, ενημερώνεται, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες ε, ε σε ό,τι φορά τις χρειάζεται πρώτερη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου πριν την προσωρινή θέση σε ισχύ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πιο λεπτομερώς αν γίνεται ποια είναι η θεσμική διαδικασία στη χώρα σας. Και σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες, ήθελα να σας ρωτήσω σε υπομοσπονδιακό επίπεδο ε, τι αρμοδιότητες έχουν οι θεσμοί, οι αυτοδιοικητικοί κάτω από το ομοσπονδιακό επίπεδο, σε επίπεδο δημοσίων προμηθειών και πώς δεσμεύονται από την όποια συμφωνία επιτευχθεί. Ναι, ευχαριστούμε. Η κυρία Σφάντ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γεια σας, ευχαριστώ κύριε Άντριος. Στην ενακτή ομιλία σα μιλήσατε για τις κοινέ αξίες Ευρώπης, Αυστραλίας. Και κάτι που είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ευρώπη και νομίζω αφορά πολύ την κοινή γνώμη όλο και περισσότερο, είναι η ανησυχία μας για τις κλιματικές αλλαγές και για το περιβάλλον γενικότερα. Εάν δούμε τι γίνεται στην Αυστραλία, ε, για μας πριν από 10 μέρες ήταν πολύ σημαντικό να δούμε την διαδήλωση, τη μαζική κινητοποίηση σε δρόμους πόλεων της Αυστραλίας πριν από 10 μέρες και μας ενέπνευσε αυτό. Η γείτον, χώρα όμως σε εσά, η Νέα Ζηλανδία, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τα Φίτζη και την Ισλανδία, την Ορβηγία για τις αλλαγές του κλίματος και την βιωσιμότητα. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προτείνει κανόνες για να ε, καταργηθούν οι επιδοτήσεις στα βλαβερά ορυκτά καύσιμα, στα επιζήμια ορυκτά καύσιμα. Στην Αυστραλία θα μπορούσατε να δείτε μια παρόμοια πρωτοβουλία, να προτείνετε κάτι παρόμοιο στις εμπορικές σας διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντάντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από την Αυστραλία. Μου άρεσε πολύ η ομιλία του εκπροσώπου της Βουλής. Με πολλά σημαντικά και επικοδομητικά στοιχεία και για μας. Αυστραλία απέφυγε με το 5G να γίνει απικία τεχνολογική της Κίνας και το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό. Θα έπρεπε να εμπνευστούμε και εμείς στην Ευρώπη. Ξέρουμε πολύ καλά τα θέματα της γεωργίας και των σχετικών συμφωνιών είναι πολύ σημαντικά και λεπτά. Για τομείς τους, όπως ξέρετε κι εσείς. Ευαίσθητος στην Ευρώπη και το ίδιο και στην Αυστραλία, τη χώρα σας. Θα ήθελα ωστόσο να τονίσω δύο πράγματα. Το σημαντικότερο για μας στη Γεωργία είναι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Θέλουμε να είναι συνδεδεμένη η γεωργιακή παραγωγή με συγκεκριμένε περιοχέ. Είναι ένα στίχημα, μια πρόκληση που ξέρουμε αντιμετωπίζουμε πριν από χρόνια και ένα μεγάλο μέρο τη γεωργία, ακόμη και πολύ μικρή κλίμακα στην Ευρώπη, ε, δεν θα υπήρχε σε διεθνέ επίπεδο και στο διεθνή ανταγωνισμό αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό και ε, προχωρούν οι σχετικέ μα διαπραγματεύσει. Κάτι άλλο που διάβασα στον ιστότοπο τη κυβέρνηση τη Αυστραλία, ο οποίο ε, πολύ καλά έχει παρουσιάσει όλε τι εμπορικέ συμφωνίε τη Αυστραλία των περασμένων ετών ή που πρόκειται να συνάψει πρόσφατα, σύντομα μάλλον, ξέρουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Και είδαμε ότι μεταξύ των προσεχών συμφωνιών μία είναι αυτή που θα υπάρξει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Brexit δεν έχει ε, πάρει κάποια μορφή ακόμα. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. Και δεν ξέρουμε αν αρχίσατε ήδη κάποια διαδικασία σύναψης συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο που θα αναθεωρεί την ε, τρέχουσα που έχετε. Ευχαριστούμε. Κάλσπροχ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για να συζητήσουμε σήμερα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το βρίσκω δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η Ευρώπη έχει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με περισσότερες από 70 χώρες, αλλά στον κατάλογο αυτό δεν εμφανίζεται η Αυστραλία. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία έχουν επιτέλους ξεκινήσει και έχουν πάρει και κάποια μορφή. Ελπίζουμε και ανυπομονούμε να έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Ζούμε σε καιρούς όπου ο προστατευτισμός και ο λαϊκισμός ε, όλο ένα και διωγγώνονται και αυξάνονται. Ο προστατευτισμός δεν μας προστατεύει ωστόσο από τίποτα. Ούτε από τον αθέμητο ανταγωνισμό, ούτε από τις κλιματικές αλλαγές. Εγώ νομίζω ότι μόνο μέσω των εμπορικών σχέσεων μπορούμε να διαμορφώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κοινό μας μέλλον. Όπως προείπαν οι συνάδελφοί μου, θα ήθελα να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και πώς μπορούμε να δούμε και την συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ και να διαμορφώσουμε και εκείνη τη συμφωνία αναλόγως για να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές. Οι εμπορικοί μα εταίροι πρέπει να είναι πραγματικοί συνεργάτε και να αντιμετωπίζουν όμω και εκείνοι με τη σειρά του τι κλιματικέ προκλήσει. Νομίζω ότι και η Ευρώπη και η Αυστραλία έχουν τεράστιε δυσκολίε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις. Ήθελα να μου πείτε λοιπόν ποια είναι η δική σα θεώρηση για τα πράγματα, Πώ το βλέπετε εσεί, Πώ θεωρείτε ότι αυτέ οι διαπραγματεύσει, αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να γίνει ένα εργαλείο αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κλίμα. Ευχαριστούμε, κυρία Χιούπνερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω για το Brexit, διότι ακούσαμε πολλά. Και αν δει κανεί και την παράδοση των εμπορικών σχέσεων με την Αυστραλία και την παράδοση που έχετε από την κοινοπολιτεία. Ξέρουμε ότι ήδη υπάρχουν κάποιε συνομιλίε Ηνωμένου Βασιλείο Αυστραλία για τι εμπορικέ σα σχέσει προσεχώ. Ξεκίνησαν πρόσφατα. Πώ βλέπετε λοιπόν τι εμπορικέ σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit, Και εκείνοι βεβαίω θα προσπαθήσουν να δώσουν μεγαλύτερο βάρο στι διμερεί εμπορικέ σχέσει με την Αυστραλία. Το βλέπετε εσείς ως ένα πιο σημαντικό σκέλος σε σχέση με τις διμερείς σχέσεις με άλλες περιοχές του κόσμου. Και ο κύριος Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία της Αυστραλίας. Χαρά μας να έχουμε τέτοιου υψηλόβαθμου προκεκλημένου και τόσο συμπαθεί. Αναφέρθηκε και προηγουμένως, περιέργως, η Αυστραλία είναι μία από τις χώρες που δεν έχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λογικό, μεν, αλλά επίσης θέλουμε τις διαπραγματεύσεις θέλουμε να προχωρήσουν και εγώ θα είμαι σκιώδης εισαγητής των σοσιαλιστών επί του θέματος. Τώρα, δύο κέρια ζητήματα θέλω να θίξω. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια συμφωνία που να είναι οικονομικά εξισυροπημένη. Η Γεωργία έχουμε ήδη πει ότι είναι ένα λεπτό ζήτημα. Πρέπει να υπάρχει επαρκής προστασία των πλέον ευαίσθητων προϊόντων μας και μετά έχουμε και το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να πάρουμε με το πλευρό μας την κοινή γνώμη, να είναι σαφές ότι μιλάμε για μια νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε ένα κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη που να είναι πιστικό η πρόσκλησή μου λοιπόν προς την Αυστραλιανή πλευρά είναι να κοιτάξετε να είναι εξυγχρονισμένη και επικαιροποιημένη η διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης στην συμφωνία. Δηλαδή θα πρέπει να επικυρωθούν μεταξύ άλλων και όλες οι βασικές συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Βλέπετε να υπάρχουν πρόπτικες να εγκριθούν από την Αυστραλία όσες δεν έχουν εγκριθεί ήδη για τον ελάχιστο μισθό ας πούμε τον κατώτατο μισθό. Και μετά για το πώ θα μπορεί να υλοποιηθεί το κεφάλαιο και οι κανόνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει ρήτρα αναθεώρηση για την ε, ισχύ των κανόνων βιώσιμη ανάπτυξη. Καλό θα ήταν να μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με του Αυστραλού φίλου ένα νέο πρότυπο για την ε, εφαρμογή και την ισχύ της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα είναι πολύ καθοριστικό αυτό για την επιτυχή διεξαγωγή των Ευχαριστούμε. Μπορείτε να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ευρείες ερωτήσεις. Σε 7 λεπτά ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους παρευρισκόμενους για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω στο μέτρο του δυνατού. Δεν ακολουθώ κάποια συγκεκριμένη σειρά. Ε, να ξεκινήσω με το Brexit. Ας μιλήσουμε για την ελέφαρα στο δωμάτιο δηλαδή. Η Αυστραλία δεν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσει ελευθερών συναλλαγών με, την, με διότι το ΕΒ Βασίλειο παραμένει μέλο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει πρώτα να γίνει το Brexit δηλαδή. Είμαστε λοιπόν πολύ πιο προχωρημένοι ε, στις διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι ακόμα και αν τελικά λάβει χώρα το Brexit, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγαλύτερος εταίρος από ότι το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, θα είναι νούμερο 3, ακόμα και αν φύγουν οι Βρετανοί, μετά την Κίνα και την Ιαπωνία. Έτσι λοιπόν, το ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει εξαιρετικά σημαντική για την Αυστραλία. Ε, γι' αυτό θέλουμε οι διαπραγματεύσει ελευθερών συναλλαγών με την Ευρώπη να προχωρήσουν. Και έχουμε φτάσει στον πέμπτο γύρο συζητήσεων. Είναι αλήθεια ότι ο Υπουργό Εμπορίου του Ενωμένου Βασιλείου ήταν πριν από μερικέ εβδομάδε στην Αυστραλία. Δεν μπορεί όμω να συμβεί οτιδήποτε από νομική πλευρά σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για την ώρα. Έχετε λοιπόν το πλεονέκτημα εσεί κατά κάποιο τρόπο στι διαπραγματεύσει. και αυτό θα το διατηρήσετε. Σε ό,τι αφορά τι τις πολυμερείς συμφωνίες τέθηκε ένα ερώτημα για τον ΠΟΕ. Εμείς δεσμευόμαστε ως Αυστραλία στην πολυμερή προσέγγιση. Γνωρίζουμε όμως ταυτόχρονα ότι ορισμένε φορές ε, οι πολυμερείς αυτές προσεγγίσεις ε, δεν μπορούν να προχωρήσουν διότι προκύπτουν συγκεκριμένα προβλήματα όπως τώρα με τον ΠΟΕ. Γι' αυτό λοιπόν προετοιμάζουμε παράλληλα και διμερείς διακανονισμούς όπου μπορούμε. Βεβαίως και εμείς δεσμευόμαστε και το πολυμερές πλαίσιο, ε, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις εκεί, ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με την Ευρώπη, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα εξακολουθούν να λειτουργούν τα πάνελ προσφυγών του ΠΟΕ ε, και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα, συμβεί, θα μπορεί να συμβεί και στο μέλλον. Κλιματική αλλαγή, βιωσιμότητα, ένα θέμα που θέθηκε από πολλούς ε, εδώ. Εμείς δεσμευόμαστε στην Αυστραλία να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ε, είμαστε υπέρ του περιβάλλοντος, θα, ε, τηρήσουμε τους στόχους του Παρισίου, των Παρισίων, ε, θα ήθελα να σας παραπέμψω ε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού μας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από ε, μία εβδομάδα περίπου. Νομίζω ότι εκεί μπορείτε να δείτε πολύ πιο λεπτομερώς ε, τις θέσεις της Αυστραλίας ε, για την κλιματική αλλαγή. Πραγματικά σας συνιστώ να ρίξετε μια ματιά σε αυτή την ομιλία, ιδιαίτερα για τα ζητήματα βιωσιμότητας, κλιματικής αλλαγής και πώς αυτό συνδέεται βέβαια ε, με τις συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών. Όλα αυτά τα ζητήματα μας πασχολούν και θα τα αντιμετωπίσουμε. Το ίδιο ισχύει και το ερώτημα του κυρίου Περέιρα που μας θύμισε τον ILO. Ε, δεν μπορώ να σας δώσω μια οριστική απάντηση για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των επαφών, αλλά είναι και, αυτό ένα θέμα που μας απασχολεί. Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, τέθηκε ένα ερώτημα για τον άνθρακα. Η αλήθεια είναι ότι οι πηγές ενέργειας οι δικές μας ήταν παρά το φυσικό αέριο και ο άνθρακας και αυτό θα εξακολουθήσει να είναι έτσι για αρκετά χρόνια. Υπάρχει αύξηση των ανανεώσιμων, πηγών ενέργεια, ε, αιωλική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι επαρκή η, η διάρκεια ζωή ε, ε, των μπαταριών αλλά βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση. Ε, το θέμα είναι πώς θα πάρει αυτή η μετάβαση. Ε, Πάντω επενδύουμε σημαντικά στις ανανεώσιμε πηγές ενέργεια στην Αυστραλία και αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ένα-δύο ακόμα ερωτήματα που τέθηκαν για τις δημόσιες προμήθειες και το επίπεδο, το υποομοσπονδιακό, το, το, το αυτοδιοικητικό. Αυτό είναι ένα ζήτημα το, βεβαίως, το, το οποίο βεβαίως θα απασχολήσει τις διαπραγματεύσεις. Ε, στο μέτρο που αυτό θα αποτελέσει μέρος του τελικού κειμένου ε, και βεβαίως δίνεται μεγάλο ενδιαφέρον στο θέμα ε, των δημοσίων προμηθειών, ιδιαίτερα στον των υπηρεσιών. Σε επίπεδο πολιτιών είναι αλήθεια ότι πολλές υπηρεσίες τις παρέχει η πολιτεία, ό,τι δηλαδή δεν προβλέπεται δεν είναι στι αρμοδιότητε τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, είναι στι αρμοδιότητε των πολιτιών και αυτό βεβαίω ε, θα αποτελέσει μέρο τη ε, συζήτηση. Έγινε αναφορά επίση στι γεωγραφικέ ενδείξει. Ε, υπάρχει ένα σχετικό κατάλογο και όλα αυτά συζητώνται. γίνεται μια δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό στην Αυστραλία. Εμεί θεωρούμε ότι μπορούμε να τα βρούμε. Ε, υπήρχαν ήδη, διακανονισμοί σε ό,τι αφορά το, το, το, κρασί, τον ίνο στην Αυστραλία. Τυπικό παράδειγμα, η σαμπάνια ε, είναι μια λέξη που δεν χρησιμοποιείται πια για το αφρόδι ίνο τον, ε, ε τον Αυστραλέζικο μετά από συμφωνία. Ε, υπάρχουν μια σειρά από προϊόντα, το τυριά, τα γνωρίζω αυτά. Ο κ. Ντάντε προφανώς έχει ενδιαφέρει ενδιαφέρει για το θέμα αυτό ως Ιταλός. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα. Να πω για το ερώτημα της κυρίας Κάλσμπρο για ε, τον προστατευτισμό και την ελεύθερες συναλλαγές. Η Αυστραλία πέρασε στη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 80 από μια φάση πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Σε ιστορικό επίπεδο εμείς ε, απαλείψαμε μια σειρά από προστατευτικά ε, μέτρα, από εμπόδια. Ανοίξαμε την αγορά μας ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι κάτι που το υποστήριξαν όλες οι πολιτικές ε, ομάδες στην χώρα μας. όχι μόνο η δική μου κόμμα, το δικό μου κόμμα το ε, αλλά και το, το εργατικό κόμμα. αν δείτε λοιπόν εκείνη την περίοδο υπήρχε μεγάλη συνένεση σε ό,τι αφορά την ανάγκη η Αυστραλία όχι μόνο να μπορεί να εμπορευθεί διεθνώς όσο καλύτερα μπορεί, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η αποτελεσματικότητα ε, θα αφορά και ε, αυτούς που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας. Ε, είμαστε μια χώρα εμπορίου, δεν είμαστε μια προστατευτική χώρα. Βεβαίως, λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα συμφέροντα του λαού μας. Εμείς δεσμευόμαστε να υπάρχει ένα σύστημα με κανόνε στο διεθνέ εμπόριο διότι θεωρούμε ότι αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ευημερία για τους Αυστραλούς, αλλά και γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Άντριους. Υπάρχει μια ακόμα επιπρόσθετη ερώτηση. Παρακαλώ, η κυρία Σάουνς. Ευχαριστώ για την απάντηση, κύριε Άντριους. Για το θέμα της κλιματικής αλλαγής αναφερθήκατε στην ομιλία του κύριου Μόρισον την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ε, του Πρωθυπουργού. Έριξα λοιπόν μια ματιά και υπάρχουν κάποιες απαντήσεις ε, σε σχέση με αυτά που είπε. Πρώτα απ' όλα γνωρίζω και ότι ο κύριος ε, Μόρισον δεν ήταν παρόν στην Σύνοδο Κορυφής για την κλιματική αλλαγή. Ε, είπατε ότι η Αυστραλία θέλει να πετύχει τους στόχους των Παρισιών, αλλά είναι από τους πιο χαμηλούς ε, για τη χώρα σας. Ο κ. Μόρισον αναφέρθηκε στην μικρή συνεισφορά της Αυστραλίας στις εκπομπές. Όμως είστε μεγάλος εξαγωγέας άνθρακα και αν το λάβουμε υπόψη μας και αυτόν, είστε υπεύθυνοι για το 20% των εκπομπών. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να απαντήσετε λίγο πιο λεπτομερό στο ερώτημα αυτό των ρηκτών καυσίμων και της επιδότησης των καυσίμων αυτών και το ρόλο που παίζει τελικά αυτό το αγαθό ε, στην παγκόσμια οικονομία και σε σχέση με την επίτευξη των στόχων. Και ο κύριος Κέλλη, μια σύντομη ερώτηση. Ε, ναι, μου αρέσει πολύ η Αυστραλία. Έχω πάει πολλές φορές εκεί. Ζουν δύο γη μου εκεί. Και θέλουμε να έχουμε μια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών μαζί σας, αλλά δεν απαντήσατε στο ερώτημά μας ε, για τη γεωργία. Υπάρχει ανησυχία ε, σε πολλούς γεωργικούς τομείς ότι το παρακάνουμε σε ό,τι αφορά τι ε, συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών ε, για τα γεωργικά προϊόντα. Και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ποιε είναι λοιπόν οι φιλοδοξίε σα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία ελευθερών συναλλαγών στον τομέα τη γεωργία. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη συμφωνία με το Μερκοσούρ, τη δική μα. Ε, θα ήθελα να ξέρω λοιπόν και εσεί ποιε είναι οι δικέ φιλοδοξίε ε, στον τομέα της γεωργίας. Ναι, να ξεκινήσω με τη γεωργία, κύριε Κέλλη. Ακούστε, προφανώς ε, οι, ε, οι γεωργοί μας, όπως και οι Ευρωπαίοι γεωργοί, θέλουν να παράγουν και να εξάγουν τα προϊόντα τους. Είναι προφανές αυτό. Και βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας. Και αυτό θα είναι και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Επίσης, θεωρούμε ότι μια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών σίγουρα περιλαμβάνει και τη γεωργία. Η γεωργία είναι ένας παράγοντας σημαντικός, αλλά είναι ένας παράγοντας. Από ευρωπαϊκή προοπτική και από πλευράς Ιρλανδίας, προφανώς ε, τα συμφέροντα των Ιρλανδών γεωργών θα είναι στην πρώτη γραμμή και εμείς από την πλευρά μας δίνουμε μεγάλη έμφαση ε, στα συμφέροντα των δικών μας γεωργών. Ε, μπορούν λοιπόν να υπάρξουν βελτιώσεις. Αν δείτε τι γίνεται παραδείγματο χάρη με τι ποσοστώσει για το βόλιο κρέα στην Ευρώπη, το βόλιο κρέας που φτάνει από την Αυστραλία έχει μειωθεί λόγω ε, της αμερικανικής αύξησης, κάτι που μας απογοητεύει. Εμείς θέλουμε να ρίξουμε να βλέπουμε μπροστά, βέβαια, να μην βλέπουμε πίσω. Δεν μπορώ να σας πω ποιο είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, βέβαια. Ε, το μόνο που μπορώ να σας πω ότι, είναι ότι εμείς ε, αντιλαμβανόμαστε ότι οι Ευρωπαίοι θα κάνουν ό,τι μπορούν για την Ευρώπη και για τους γεωργούς της το ίδιο θα κάνουμε και εμείς για την Αυστραλία, για τους Αυστραλούς και για τους Αυστραλούς γεωργούς. Στον τομέα του Βόλου Κρέατος, παραδείγματο χάρη, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει πλημμυρίσει την αγορά της Ευρώπης ε, το βόλιο κρέας από την Αυστραλία. Είναι πολύ μικρό το μεριδιό μας, ε, εάν δείτε τα συνολικά, τις συνολικές ποσότητες. Το ζήτημα είναι κατά πόσο και οι δύο πλευρές μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία που σε γενικές γραμμές ε, θα προωθήσει το, εμπόδιο, το εμπόριο μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από δική σας προοπτική, βέβαια εσείς θέλετε να προστατεύσετε κάποιες πτυχές ε, των γεωργικών σας προϊόντων και της παραγωγής σας. Ε, τελικά αυτό θα κριθεί στη διαπραγμάτευση. Εάν όμως ε, εμείς προσέλθουμε στις διαπραγματεύσει αυτές καλή την πίστη, ε, νομίζω πως είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας για την διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ δυστυχώς να σας πω κάτι πιο λεπτομερές επ' αυτού, διότι ε, αυτή η λεπτομερής απάντηση θα την έχουμε μπροστά μας όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Ε, κυρία Τσάουνς, ε, σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό μας είναι η άποψη της Αυστραλίας. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικούς στόχους σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Παρισίων, είναι όμως στόχοι που είναι αντικείμενο συμφωνίας, ευρεία συμφωνίας. Ε, στην Αυστραλία υπάρχει μεγάλη συνένεση από αυτών των στόχων. Έχουμε πολλά πολιτικά κόμματα, αλλά όλοι συμφωνούν να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Τώρα για τον άνθρακα, ναι, είναι αλήθεια ότι εξάγουμε άνθρακα. Όμως, οι εξαγωγές μας άνθρακα είναι ε, καλύτερες, είναι μικρότερες από ό,τι από άλλες χώρες του κόσμου. Ε, είμαστε στη μεταβατική φάση. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε ότι εγκαταλείπουμε τον άνθρακα ή το φυσικό αέριο. Δεν έχουμε πυρηνική ενέργεια όπως έχουν διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ε, γίνεται μια συζήτηση και για την πυρηνική ενέργεια στην ε, Ευρώπη. Έχουμε τις μεγαλύτερες πηγές ουρανίου στον κόσμο, αλλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι γνωρίζουμε ότι είναι ευαίσθητα τα ζητήματα αυτά, γνωρίζουμε ότι γίνεται προσπάθεια ε, για το θέμα αυτό σε όλο τον κόσμο ε, και εμάς μας ανησυχεί το θέμα με βάση τη δική μας εμπειρία, τη δική μας ιστορία ε, δεν παραβλέπουμε τα ζητήματα που θέσατε, μας τα θέτουν και άλλοι αλλού. Είναι μια συζήτηση που βρίσκεται να εξελίξει και θα συνεχιστεί και στην οποία συζήτηση αυτή θα συμμετάσχουμε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ο Peter Birds από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Είναι ο ειδικό τη διαπραγματεύση με την Αυστραλία και θα μας πει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού βρισκόμαστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε Λάγκε. Ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων εδώ. Τις απόψεις και από το Κοινοβούλιο και από την Αυστραλία. Και χθε στην αντιπροσωπεία είχαμε ανταλλαγή απόψεων πολύ ε, καλή και επίκαιρη. Ο Επίτροπος Χόγκαν παρουσίασε επίσης τις απόψεις του την περασμένη Δευτέρα για την εμπορική πολιτική και είχαμε και την ομιλία της ε, Πρόεδρο της Επιτροπής Φόντερ Λάιεν και ε, κάποια συμπεράσματα. Είχαμε, έχουμε σημαντική εμπορική σχέση παρά τη μεγάλη απόσταση. Το όγκος του εμπορίου αυξάνεται, είμαστε κοντά στα 50 δις ευρώ κάθε χρόνο και μπορούμε να βελτιώσουμε το νούμερο αυτό, έξω και οι διαπραγματεύσεις για οικονομικούς αλλά και γεωπολιτικούς λόγους ε, κατέρωθεν. Εμείς, όπως επιβεβαιώθηκε σήμερα, έχουμε τις ίδιες αξίες, τους ίδιους στόχους στο εμπόριο. Είμαστε δεσμευμένοι να έχουμε ε, ένα σύστημα πολυμερές στο εμπόριο, βασισμένο σε κανόνες. Ε, είχαμε, έχουμε πέρα από τις διαπραγματεύσεις συνεχιζόμενες και συνεχή διάλογο για θέματα εμπορίου όπου συζητούμε ευρύ φάσμα θεμάτων από θέματα ε, που είναι προβλήματα διμερή μέχρι θέματα του ΠΟΕ. Ε, προχωρούμε με καλό ρυθμό. Δύο μήνες μετά την ε, αποδοχή της εντολής αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις. Η εντολή πήρε κάποιο χρόνο και στο Συμβούλιο και επειδή ε, πέρασε πολύ χρόνος για να προετοιμάσουμε τις διαπραγματεύσεις με τους Αυστραλούς εταίρους με ένα προπαρασκευαστικό έγγραφο που κατέγραφε τις κοινέ μας φιλοδοξίες από τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ε, ήταν μια σωστή ε, επένδυση αυτή γιατί διευκρινίζει στόχους και εξοικονομεί χρόνο από τις καθ' αυτό διαπραγματεύσεις. Ο τέταρτος διαπραγματευτικός γύρος έγινε στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο και τώρα προχωρούμε προς τον το 14 14-18 Οκτωβρίου στην Κανμπέρα και έχουμε καλή βάση σε όλους τους τομείς των διαπραγματεύσεων για να συνεχίσουμε. Βέβαια, τα εύκολα τα, προχωρού, τα προσπερνάμε γρήγορα, αλλά θα έχουμε και αρκετά δύσκολα να δούμε με τη συμμετοχή του το Ευρωπαϊκό και το Αυστραλιανό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσουν. Έχουμε φιλόδοξες προσδοκίες. Η διαπραγματευτική εντολή ζητεί από την Κομισιόν να διαπραγματευτεί μια ΣΕΣ, μια Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών φιλόδοξη. Υπάρχουν οι προθέσεις και στο παρασκευαστικό έγγραφο και στην εντολή και Έχουμε τον τομέα της γεωργίας, ευαίσθητος τομέας όπως είπαμε και σήμερα. Κάποια θέματα στο ε, χαρτοφυλάκιο της γεωργίας πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και ως προς αυτό καταστήσαμε σαφές στην Αυστραλία ότι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων είναι κάτι που θεωρεί πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η νέα κυβέρνηση ελπίζω, επήρε το ένα σημαντικό βήμα μέσα Αυγούστου για να δημοσιεύσει τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρώπης. Ε, καθυστέρησε κάποιους μήνες, αλλά τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανταλλαγή των ε, προσφορών εις ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά που θέλουμε να ολοκληρώσουμε πριν από τον πέμπτο γύρο. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως επενδύσεις, ε, δημόσιες συμβάσεις, ε, ε, αυτά ακολουθούν και τώρα ο τομέας των υπηρεσιών αυξάνεται. Είναι πολύ σημαντικός ο τομέας αυτός, δεδομένης παγκοσμιοποίησης και επειδή πρόκειται για οικονομίες τους αντίποδες, καλό είναι να έχουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο για τις υπηρεσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στις ε, σχέσεις μας. Επίσης σημειώσαμε με ικανοποίηση ότι η Αυστραλία ε, προσχώρησε στην Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις ε, του ΠΟΕ πριν από το καλοκαίρι. Αυτό είναι καλό και θα βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις μας με βάση τη διαφάνεια της μη διακρίσης. Σε αυτό το τομέα ήδη έχουν γίνει σημαντικές ε, πρόοδοι ε, στους τελευταίους γύρους. Ε, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική. Εδώ ακούσαμε τις απόψεις και προσδοκίες από εδώ. Θέλουμε το εμπόριο να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη, κλιματικές δράσεις. Στις διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία θα υπάρξουν προθέσεις για να υπάρξουν αποτελέσματα εδώ. Επίσης οι προτάσεις μας για αυξημένο εμπόριο παράλληλα με την ε, κλιματική αλλαγή, της, ε, την συμμόρφωση προς τις αρχές της ILO, ε, όλα αυτά έχουν διατυπωθεί. Ηρίστο εμπαρόδο, εσωτερικά κάνουμε και μία μελέτη επιπτώσεων για την εφικτότητα είναι μια μελέτη που γίνεται από ανεξάρτητο ανάδοχο ε, και εξετάζει την ΣΕΣΕ που διαπραγματευόμαστε ως προς τους ε, περιβαλλοντικούς ε, και κοινωνικούς αντίκτυπους που μπορεί αυτή να έχει. Η τελική έκθεση θα είναι στα χέρια μας στο τέλος του έτους. Επίσης, ε, ε, ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95% των επαγγελματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να τους έχουμε υπόψη λοιπόν γιατί θα πρέπει το εμπόριο να εξυπηρετεί όχι μόνο τις μεγάλες αλλά για τις μικρές επιχειρήσεις και εκείνες πρέπει να δρέψουν ωφέλη από αυτήν τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Έτσι λοιπόν όλα αυτά είναι σημαντικά για τις διμερείς μας σχέσεις και αυτό είναι να, οι διαπραγματεύσεις είναι, ε, δίνει αν θέλετε ένα μήνυμα και για τις ε, απόψεις που έχουμε σε σχέση με το ε, δίκαιο εμπόριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, ο εισηγητής μας, ο Ντανιέλ Κασπάρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων. Σήμερα είχα την εντύπωση ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής φαίνεται να βλέπει θετικά τις συνομιλίες αυτές. Σίγουρα πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ για την ενημέρωση από Αυστραλιανής πλευράς. Είναι καλό για να καταλάβουμε καλύτερα τα θέματα και ε, τα σχόλια των συναδέλφων ήταν πολύ θετικά. Είχαμε μια καλή ακρόαση και μελέτες επίσης σε σχέση με το εμπόριο και το περιβάλλον. Κάποιοι ανέφεραν το θέμα αυτό, ίσως μπορούμε να το θέσουμε σε κάποια μελλοντική ημερήσια διάταξη, γιατί θα βοηθήσει και τη συμφωνία με την Αυστραλία. Το, εμπόδιο, το εμπόριο επηρεάζει θετικά αλλά και αρνητικά το περιβάλλον. Ίσως θα πρέπει να δούμε ξανά το θέμα αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να συνεχιστούν οι επιτυχείς διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Κλείνει η συζήτηση εδώ. Εύχομαι στους Αυστραλούς ε, προσκεκλημένους να κερδίσει η Αυστραλία τον αγώνα ράγμπι του Σαββάτου και ε, σας εύχομαι καλό ταξίδι και ό,τι το καλύτερο. So, Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Για να είμαι εντελώ ειλικρινή, ψάχνω τον εισηγητή και δεν τον βλέπω. Τον εισηγητή για το Βιετνάμ. Α, Okay. Okay. Now we... Ωραία. Περνάμε σε μια άλλη σημαντική συμφωνία, κάπως πιο συγκεκριμένη. Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και συμφωνία για τις διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ. Δύο συζητήσεις θα έχουμε και θα έχουμε και ένα κοινό ψήφισμα. θα έχουμε 4 και 5 για, την, ε, για τις ελεύθερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα για τις ε, διαπραγματεύσεις, για τις επενδύσεις, συγγνώμη. Έχουν μεταφραστεί, έχουν διατεθεί τα κείμενα από το Ευρωκοινοβούλιο και σκοπός μας τώρα είναι να αξιολογήσουμε τη συμφωνία και για την κύρωση και σε αυτό το πλαίσιο θα οργανώσουμε και επίσκεψη στο Βιετνάμ τέλη Οκτωβρίου. Θα δούμε τις εξελίξεις εκεί. και πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία για την τελική επεξεργασία των συμφωνιών εδώ στο Κοινοβούλιο. Μετά θα υπάρξει προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών μετά την επιστροφή της αντιπροσωπείας της Βρυξέλλες. Αυτή είναι η δική μου η εισαγωγή. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Φράγκο, που αντικαθιστά τον εισηγητή, τον κύριο Ζάχραντιλ. Όμως ούτε εκείνο είναι εδώ. Το σημειώνουμε στο αποσιολόγιο. Ο κύριος Μπέτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Λάγκε. Μπορώ να μιλήσω και για τον εισηγητή, αν θέλετε. Καλά. Αγαπητοί βουλευτέ, χαίρομαι που μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Επιτροπή σα και κατά σύμπτωση αύριο κλείνουμε μία επέτειο το είχαμε συζητήσει πάλι στην Επιτροπή σα πριν από ένα χρόνο, οπότε ευκαιρία να σα ενημερώσω για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και η, συμφων... η συνάδελφό μου η Μαρία θα σα ενημερώσει για τι επενδύσει. Την Συμφωνία Προστασία των Επενδύσεων. Όπω είπατε, Πρόεδρε, οι υπογραφέ και των δύο συμφωνιών έλαβαν χώρα στι 30 Ιουνίου. Ορόσημο για την όλη διαδικασία. Πήρα και κάποια χρόνια βέβαια μέχρι να ολοκληρωθούν οι συμφωνίε και σκοπό έχουν να συμπληρώσουν το πλαίσιο των σχέσεων που έχουμε με το Βιετνάμ. Ήδη έχουμε συμφωνία εταιρική σχέση και σύνδεση. Συνεργασία, μάλλον, συγγνώμη. Οπότε τώρα θα έχουμε περαιτέρω εμπορικέ και επενδυτικέ σχέσει και δεσμού. Πολύ καλό δείγμα, όχι μόνο για την διμερή εμβάθυνση των ε, αμοιβαίων υποσχέσεών μα, αλλά είναι και ένα μήνυμα προ τον υπόλοιπο κόσμο ότι προχωρούμε. Θέλουμε ένα εμπόριο το οποίο να βασίζεται σε διεθνείς σχέσεις και αυτό θέλει να τονώσει και την παρουσία μας στην Ασία. Έχουμε τώρα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μόνο με την Κορέα και την Ιαπωνία προς στιγμή. Αν όλα πάνε καλά, γρήγορα θα έχουμε και την Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Οπότε έτσι ε, ερχόμαστε σε επαφή με πολλά μέλη της ΑΖΕΑΝ. Η Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ θα είναι ακριβώς ε, η πρώτη κρίκη μια τέτοιας ε, διαδικασίας σύνδεση. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μας φέρνει σε καλύτερη συνεργασία ε, και με ανταγωνιστές μας, τρίτες χώρες που ήδη έχουν Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με το Βιετνάμ. Θέλουμε να τις προλάβουμε και να τις ξεπεράσουμε στον αγώνα δρόμου. Να τονίσω κάποια τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η πιο φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που έχει ποτέ αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτη χώρα. Θα απαλείψει όλου του δασμού, όλου του εξαγωγικού δασμού, μάλλον μεγάλο αριθμό των εξαγωγικών δασμών. Η γεωργία, κτηνοτρόφια και οι εταιρείε θα εποφεληθούν από 196 προστατευόμενε ενδείξει μέσω τη ε, ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και το Βιετνάμ ω προ τα φυτο-υγειονομικά και υγειονομικά μέτρα θα αναγνωρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ω μία απόσταση. Επίση, για συμβάσει και προμήθειε θα μπορεί να υπάρξει, διαφανή διαδικασία. Θα απομακρυνθούν οι μη δασμολογικοί φραγμοί. Και το Βιετνάμ θα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα στι διμερεί μα σχέσει. Επίση, έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τις προδιαγραφές για πολλές υπηρεσίες, περιβαλλοντικές και ούτω καθεξής. Επίσης, οι κανόνες ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Βιετνάμ θα είναι ίσες με τις υπόλοιπες ε, και δεν θα υπάρχουν επιδοτήσεις για να μην υπάρχει άδικη διοικητική μεταχείριση κατά των ευρωπαϊκών εταιριών καθώς και προστασία της πνευματική ιδιοκτησίας με ένα ανάλογο ισχυρό κεφάλαιο. Έχουμε βεβαίως και δείκτες αξιολόγηση, συγκριτικής για αυτή τη συμφωνία καθώς και για τις υπόλοιπες χώρες της ΑΖΕΑΝ. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό κεφάλαιο TST και βλέπουμε βεβαίως και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, την περιβαλλοντική προστασία Όλα αυτά αναφέρονται στο προήμιο της συμφωνίας. Όλα όσα, όλα όσα αφορούν το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με εργασιακά πρότυπα, περιβαλλοντικούς κανόνες, ένα μηχανισμό επιλύσης των διαφορών και τη θέσπιση συμβουλευτικών ομάδων ε, εσωτερικώς. Για μια αναπτυσσόμενη χώρα όπως το Βιετνάμ, πρώτη φορά Έχουμε ένα κεφάλαιο με διατάξεις TST παρόμοιες με αυτές που είχαμε σε συμφωνίες με ανεπτυγμένες χώρες όπως ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Θα πρέπει κάποια στιγμή το Βιετνάμ να ετοιμαστεί για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από όλες τις διατάξεις TST και βεβαίως το Βιετνάμ ακόμα δεν έχει κυρώσει τρεις από τις βασικές συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού εργασία, Την ε, σύμβαση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις κυρίως και έχουμε και έναν οδικό χάρτη για τις υπόλοιπες δύο που απομένουν, όπως την Συμφωνία Σύνδεσης. Το Βιετνάμ πάντως έχει εγκρίνει μια οικειοθελή συμφωνία για την ε, προστασία των δασών, την ε, καταπολέμηση της αποξύλωσης. Και είναι η χώρα της Ασίας που έχει σεβαστεί τις περισσότερες ε, συμβατικές μας υποχρεώσεις στη συμφωνία της, έχει λάβει υπόψη. Για, τις για, για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα έχουμε συζητήσει με το Βιετνάμ Έχουμε καθορίσει τα πράγματα με βάση την προηγούμενη συμφωνία σύνδεση και συνεργασία, οπότε επαναλαμβάνονται κάποιε σχετικέ διατάξει, μεταξύ των οποίων μερική ή ε, ολοσχερή αναστολή τμήματων τη συμφωνία. Όπω είπε ο πρόεδρο, κάποιοι από εσά θα επισκεφτείτε τον Βιετνάμ στο τέλο του μήνα, οπότε είμαι βέβαιο ότι θα περάσετε ωραία και ότι θα σα φιλοξενήσουν πολύ ευχάριστα και ελπίζω ότι η Εθνοσυνέλευση που συνεδριάζει αυτό και τον επόμενο μήνα, θα έχει καλύτερα και πιο ευχάριστα νέα για τη διαδικασία υλοποίηση κύρωση και έγκριση των όσων πρέπει να ενταχθούν στον εργατικό κώδικα, στο εργατικό δίκαιο. Είναι υποχρεώσει που έχει αναλάβει το Βιετνάμ στα πλαίσια τη σύνδεση του με το Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασία. Χαρά μου λοιπόν να συνεργαστώ με τα μέλη τη Επιτροπή σα και ανυπομονώ για τη γρήγορη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Το Βιετνάμ, λοιπόν, θα συζητήσει την ε, αναθεώρηση του εργατικού, του εργατικού δικαίου τις συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας που πρέπει να ενταχθούν ε, στην ομοθεσία της χώρας και βεβαίως για να προχωρήσει η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Οι συλλογικέ διαπραγματεύσει είναι ένα σαφέ βήμα. Για να υπάρξει πραγματικά μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου. Οπότε ελπίζουμε αυτό να προχωρήσει για να έχουμε μια σαφέστερη προοπτική. Και τώρα ο λόγος στον συνάδελφο που αντικαθιστά τον εισηγητή μας, κύριε Φράγκο, για πέντε λεπτά. Gentlemen, I'm here today in step Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω έρθει για να αντικαταστήσω τον ε, συναδελφό μας, τον ε, κύριο Ζαχραντήλ, για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Βιετνάμ, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα, οπότε δεχτείτε τη συγγνώμη του. Θα σας διαβάσω τις σημειώσεις του και να σας θυμίσω ότι έχει προηγηθεί. Οι διμερείς σχέσεις και διπλωματεύσεις με το Βιετνάμ ξεκίνησαν το 2012 και ολοκληρώθηκαν σε πολιτικό επίπεδο το Δεκέμβριο του 2015. Η καθυστέρηση αυτή, αν μπορώ να πω, έχει να κάνει με τον διαχωρισμό εξουσιών. και τις προεδρικές εκλογές στη Σιγκαπούρη που οδήγησαν τελικά σε δύο ξεχωριστές συμφωνίες. Τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και τη Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων. Κατά δεύτερον, η καθυστέρηση έχει να κάνει και με τις εσωτερικές μας διαδικασίες, μεταφράσεις, ε, και το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να έχουμε συγκατάθεση ε, στην προηγούμενη φοιτεία. Με συγχωρείτε για τα αγγλικά, δεν είναι τόσο καλά. Ευχαριστώ. Η φτωρινή καθυστέρηση δεν είναι αποδεκτή, αλλά εάν δεν καταφέρουμε να φέρουμε σε ισχύ όσα έχουμε υποσχεθεί μέσω της συμφωνίας, δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Πώς θα μας βλέπουν οι εταίροι μας, ε, τι θα πιστέψουν για μας. Πρέπει να προχωρήσουμε με τη διαδικασία κυρίως όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Υπάρχουν οικονομικά εφέλη που τα αναμένουν και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Και επανειλημμένως το έχω πει, οι εμπορικές μας πολιτικές δεν έχουν μόνο την, να κάνουν με την αύξηση του ΑΕΠ, αλλά και μοναδικές ευρωπαϊκές αξίες. Αυτή ακριβώς η συμφωνία είναι ένα μοντέλο για να προωθήσουμε τις ε, ε μας, δίνοντας όθηση στις μεταρρυθμίσεις με, την, με το κεφάλαιο για τις εμπορικές σχέσεις θέλουμε να βελτιώσουμε το ε, τοπικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, καθώς και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Με υποσχέσεις ότι θα γίνουν συγκεκριμένα βήματα, υποσχέσεις που έχουν δώσει οι αρχές του Βιετνάμ. Οι επενδύσεις είναι ένας τρόπος για να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες και τα πρότυπα ε, στα διεθνή επίπεδα και στα ευρωπαϊκά. Ε, οι υποσχέσεις για μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου έχουν να κάνουν με την κατάργηση της παιδικής εργασίας ή την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, της ε, πωλήσης στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει πλήρη προσχώρηση στι συμβάσει του ε, Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασία. Έχουμε έναν οδικό χάρτη, υποσχέσει και πρέπει να δούμε και αποτελέσματα. Τίποτα βέβαια δεν μπορεί να είναι απόλυτα τέλειο, αλλά παρόλο που πρέπει περισσότερα να γίνουν, είναι μια διαδικασία όπου η εμπορική συμφωνία σκοπό έχει να βοηθήσει ε, τι μεταρρυθμίσει σε ταχύ ρυθμό, παρά να προβλέψει μια σειρά από προποθέσει. Ε, Ελπίζουμε λοιπόν αυτό να βελτιώσει το κλίμα των επενδύσεών μα. Συνάδελφοι, ελπίζω ότι μπορώ να υπολογίζω στη στήριξή σα και ότι μπορούμε να φέρουμε σε αίσιο πέρα ε, την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχουν οι σκιώδει συγγητέ για δύο λεπτά. Ο καθένα από το ΕΠΠ, ο κ. Χάνσεν από το ΕΛΚ. Δεν με έχουν ακόμη επιβεβαιώσει ο σκιώδη συγγητή, αλλά θα πάρω το λόγο παρόλα αυτά στο όνομα τη πολιτική μου ομάδα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σωστά ανέφερε ότι είναι η πρώτη και πιο φιλόδοξη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που ολοκληρώνουμε με μια αναπτυσσόμενη χώρα, αναδιόμενη χώρα, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, σημαντικό σημείο αυτό, πρέπει να το τονίσουμε. Ε, θα απαλληθούν 99% των δασμών, πολύ υψηλό ποσοστό. Ταυτόχρονα ε, μια, φορά, μια σειρά από αριθμιστικά εμπόδια θα απαλληφθούν και 169 γεωγραφικές ενδείξεις δικές μας θα προστατεύονται ε, με βάση τις διπραγματεύσεις αυτές. Ε, είναι το δεύτερο βήμα μας στην ασιατική αγορά. Για γεωπολιτικούς λόγους είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι σχέσεις μας με την με το ασιατικό μπλοκ. Πολύ σωστά είπε η Κομισιόν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και στο κεφάλαιο του, που αφορά στο TST, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την, την επικύρωση της σύμβασης του ILO για τις συλλογικέ συμβάσεις και βεβαίως παραμένουν ακόμα, εκκρεμούν ακόμα δύο συμβάσεις του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, για τι γεωγραφικέ ενδείξει όμω θα ήθελα να μου πείτε κάτι περισσότερο, περισσότερες εξηγήσεις περιπτώσει, για το πώ προχωράει η διαδικασία με τι γεωγραφικέ ενδείξει με το Βιετνάμ, για την αναγνώριση δηλαδή και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεών μα και δεύτερον, οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο για το Βιετνάμ μετά την Κίνα και το δεύτερο, η δεύτερη αγορά εξαγωγών ε, μετά τις ΗΠΑ στην Ευρώπη ε, πώς ε, θα εξασφαλίσουμε ότι το Βιετνάμ δεν θα γίνει πίσω πόρτα των Κινέζων για να μπορέσει να εξάγουν προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτή είναι η πρώτη συνολική σφαιρική συμφωνία, συμφωνία ελευθερών συναλλαγών με μια αναπτυσσόμενη χώρα. Ε, πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει μια γεωπολιτική διάσταση ε, έντονη. Το Βιετνάμ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζουμε από τις συζητήσεις μας ότι υπάρχει μεγάλη πτυτικότητα αυτή τη στιγμή, μεγάλη αστάθεια ε, στο εμπορικό κλίμα παγκοσμίω. Ε, για το Βιετνάμ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εταίρος αξιόπιστος και σταθερός σε έναν αβέβαιο κόσμο. Ε, είναι πολύ καλό ότι υπάρχει μια συμφωνία και στον τομέα της δασοκομείας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει καλή πρόθεση. Θα πρέπει εμείς να τονίσουμε τα δυνατά μας σημεία κατά τη γνώμη μου. Εμείς ε, προσφέρουμε μια ισχυρή και σταθερή σχέση. Πρόσβαση στη μεγαλύτερη, στο μεγαλύτερο ε, μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Και αυτό έχει ένα κόστο. Πρέπει να είναι σαφέ δηλαδή για του Βιετναμέζου ποιε είναι οι προποθέσει για να έχουν πρόσβαση στην αγορά μα. Ε, υπάρχουν τα οι παραβαλλοντικέ ε, ε απαιτήσει που έχουμε, οι απαιτήσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλου του εταίρου μα και ιδιαίτερα για τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε στα πλαίσια του GSP, θέλουμε επικύρωση και εφαρμογή και παρακολούθηση ε, των συμβάσεων αυτών. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι λιγότερο ε, από αυτά που ζητάμε από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα από τις αναδυόμενες οικονομίες όπως το Βιετνάμ. Ε, διότι αλλιώς είναι σαν να υπονομεύουμε τη δική μας, τη δική μας εμπορική πολιτική. Σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο πλαίσιο πολύ σύντομα, σας το υπόσχομαι. Είχαμε μια συμφωνία συνεργασία και εταιρική σχέση από το 2016 με έναν διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2012 και μετά υπάρχει ένας διάλογος για τη βιώσιμη ανάπτυξη τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια του FTA. Από το 2012 κάθε χρόνο ε, υπάρχουν πιο πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές στο Βιετνάμ. Το το 2019 Human Rights Watch μας λέει ότι είναι όλο και χειρότερος ο απολογισμός ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μιας και ε, υπάρχουν άνθρωποι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη φυλακή, δρα, δρακόντιοι νόμοι που ε, απειλούν το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Η Διεθνής Αμνηστία λέει ότι η πολιτική κρατούμενη, η κρατούμενη συνείδηση έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς σε αυτήν την ε, επιτροπή. Η κατάσταση με ανθρώπινα δικαιωμάτων στο Βιετνάμ είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Αναγνωρίζω ότι βεβαίω έχουμε κάποια θετικά βήματα για τα εργασιακά δικαιώματα. Είχαμε την επικύρωση του 1998. Είναι όμω πολύ σημαντικό, διότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακούστε, όλοι τα ίδια δικαιώματα έχουμε όμω, λέει ο πρόεδρο. Ήθελα να πω ακόμα κάτι. Το, το δεν είναι τίποτα χωρίς το 87. Η κυρία η Κάριν έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και βεβαίω αναμένουμε την μονησία τη περαιτέρω συζητήση. Θα συμμετάσχω και στην αντιπροσωπεία του Βιετνάμ. Ε, εγώ πιστεύω ότι η εμπορική συμφωνία είναι ένας τρόπος ε, δημιουργίας ε, συμπράξεων, εταιρικών σχέσεων, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, να γίνουν συζητήσεις και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι και ένα εργαλείο για να τονίσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, ε, πολιτικές ελευθερίες, ε, ε ελευθερία λόγου και τα λοιπά. Χαίρομαι που το Βιετνάμ έχει κάνει κάποια βήματα για να επικυρώσει σημαντικές συμβάσεις. Το ζήτημα όμως είναι τι μπορούμε να πούμε τελικά για τη δυνατότητα εφαρμογής, ε, υλοποίησης. Θα χρειαστεί τεχνική συνδρομή, θα χρειαστούν άλλα πράγματα για να σπρώξουμε λίγο το Βιετνάμ προς την θετική κατεύθυνση. Ε, λίγο μαστίχιο και λίγο καρότο. Ε, ιδιαίτερα στο σύστημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Σφόρτσα για τους πρασίνους. Είμαι σκιώδης ε, και για την ΔΕΒΕ. Το Βιετνάμ αναπτύχθηκε οικονομικά πολύ γρήγορα, εμπορικά επίσης, καταπολέμησε έτσι και τη φτώχεια. Το Βιετνάμ ακόμα είναι μονοκομματικό κράτος. Αναφέρατε πριν από ένα χρόνο ε, ένα ψήφισμα που πέρασε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ και πριν από μία εβδομάδα ακούσαμε ότι δεν βελτιώθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντίθετα επιδεινώθηκαν ε, κατά την περίοδο αυτή. Τώρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ως μοχλό για να διασφαλίσουμε βελτίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο περιβάλλον κλπ. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο πριν υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει η αλλαγή αφού υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία. Γιατί ιδιαίτερα με τα, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιδεινώνεται θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε ε, μια ε, υποχώρηση από τη δική μας την πλευρά. Επίση, η Σύμβαση 87 της ΑΕΛΟ έχει ε, υπογραφεί, αλλά ο ποινικό κώδικας της χώρας έχει ε, προβληματικά σημεία σχετικά με το δικαίωμα του συναθρίζεστε, ειρηνικές συναθρήσεις κλπ ή τη διακυβέρνηση, πολιτικά δικαιώματα που δεν, ε, δεν, δεν υπάρχουν. Πώς μπορεί λοιπόν η εμπορική πολιτική να παίξει ρόλο με, την, με το Μερκοσούρ είδαμε ότι δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τακτική του μαστίγιου και του καρότου. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση και αν δεν μπορούμε τώρα να ε, χρησιμοποιήσουμε τις συμφωνίες ως μοχλό για πριν από την ε, κύρωση της συμφωνίας για να ε, επιτύχουμε κάποιες βελτιώσεις, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε μετά. Και με την Ιαπωνία το είδαμε ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας ε, ε, αισθάνονται όλοι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο κύριος Λαντσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέμε για προστασία του περιβάλλοντος, για ανθρώπινα δικαιώματα, για κυκλική οικονομία, για προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, όμως στην πράξη. Ποιες είναι οι δράσεις που θα προβλεφθούν για να παρακολουθήσουμε κατά πόσο αυτές οι υποσχέσεις τηρούνται στην εμπορική συμφωνία. Και εν τέλει, εάν δεν τηρηθούν, ποιες είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που θα έχουν, ε, διατάξεις που θα έχουν προβλεφθεί στην εμπορική συμφωνία, ώστε οι εταίροι μας να υποχρεωθούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Πολλά ωραία λόγια ακούμε, αλλά στην πράξη όταν υπάρχει ανάγκη δράσης, βλέπουμε ότι έχουμε έναν τέρο απέναντί μας κάπως ε, μεταβαλλόμενο στη στάση, για να το πω απλώς. Ευχαριστούμε για την ΚΟΕ. Ο κύριος Σόλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή για την ενημέρωση ε, και εκ μέρους του σκιώδους εισηγητού μας. Πρέπει να πω ότι βλέπουμε να υπάρχει μια σχετική βελτίωση στα εργασιακά δικαιώματα και διάθεση μεταρρύθμισης στη χώρα. Τον Οκτώβριο ανακοινώθηκε ότι θα συζητηθεί η μεταρρύθμιση του εργατικού κώδικα, στην, του εργατικού δικαίου στην Βουλή της χώρας και να γνωρίζουμε ότι η σύμβαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας του 1998 είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να περάσει. Και στην περίπτωση του Βιετνάμ, ε, πρέπει να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα. Για τις ε, διατάξεις TST ε, μας είπατε ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό κεφάλαιο. Αλλά είναι δεσμευτικές αυτές οι διατάξεις Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε ε, και να δούμε με τους Βιετναμέζους εταίρους, με τις εταιρείες, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά πόσον μπορούμε να φέρουμε τους Βιετναμέζους πιο κοντά στις αξίες μας. και να φροντίσουμε η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών να είναι εργαλείο που να βελτιώσει τις συνθήκες και τις οικονομικές αλλά και τις κοινωνικές. Και σημαντικό είναι να συμπεριλάβουμε στη συμφωνία μια ρήτρα προστασίας για τις μειονότητες και τις κοινότητες που μπορεί να ε, απειλούνται. Εδώ πρέπει να αναλάβουμε αυτή την υποχρέωση απέναντι στους εταίρους μας. Έχουμε ευθύνη, διότι λέω ναι, οι διαπραγματεύσεις έχουν φέρει ένα συγκεκριμένο βαθμό σύγκλησης, αλλά πρέπει να πάμε παραπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως ξέρετε, τρεις επιτροπές θέλουν να γνωμοδοτήσουν σχετικά. Και για την Επιτροπή Αλίας έχουμε τον κύριο Μπαρτόλη μαζί μας για τα σχόλιά του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Συνάδελφοι, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε. Για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό όπου είμαι εισηγητή εκ μέρου τη Επιτροπή Αλία. Κατά την άποψή μου, είναι μια καλή ευκαιρία για τον αλληλευτικό μα τομέα η συμφωνία αυτή και είναι θετικό το γεγονό ότι η συμφωνία αναγνωρίζει τη σημασία τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την προώθηση της ε, βιώσιμη θετοκαλλιέργειας. Θεωρώ θετικό ότι οι δύο πλευρές έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για να καταπολεμήσουν την αδήλωτη, άναρχη και παρανομιαλία κάτι που είναι σίγουρα μία καλή είδηση. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ θα ε, ε, λάβει υπόψη της ε, αυτή τη δέσμευση που ζητάται και από την Επιτροπή Προστασίας των Ιδάτων στον, κεντρικό και δυτικό ειρηνικό ωκεανό. Είναι βάσει της συστάσεις, των συστάσεών του. Επίσης θα πρέπει να προστατεύσουμε τα οικονομικά μας συμφέροντα ε, και της ε, αλληλευτικής μας βιομηχανίας στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Πρέπει να υπάρχει βιώσιμη διαχείριση των αλληλευτικών και πόρων και των ίδιων των νυχθείων. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε και τη δυσκολία του Βιετνάμ να υλοποιήσει στην εθνική νομοθεσία διατάξεις για τα ανηλία νέων μεθόδων ε, παρακολούθησης και ελέγχου της παράνομης αλίας. Αυτές τις δυσκολίες τις, έχουν, έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τουλάχιστον δύο σημεία. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσω τη διάθεση του Βιετνάμ να αντιμετωπίσει την, ε, τις διαστάσει διαστάσεις του στόλου του, ώστε να πάυσει και η παράνομη αναρχική αδήλωτη αλία δεν μπορεί παρά να αποτελεί μέρος ε, μιας άσκησης παρακολούθησης μια τέτοια κίνηση από το Βιετνάμ. Μια άσκηση που θα πρέπει να είναι συνεχής και με διεξοδικούς ελέγχους για να μπορούμε επικοδομητικά να βλέπουμε αν οι συνδυασμένε κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν. Τέλος, είναι σημαντικό στα πλαίσια της συμφωνίας να υπάρχουν εγγύησεις ώστε η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά μας να συνοδεύεται από συγκεκριμένες διασφαλίσεις. Χρειάζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου με περιόδους ε, παρακολούθησης. Θα πρέπει να είναι σαφή η δυνατότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωση να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει για να σηκώσει κόκκινη κάρτα εάν χρειαστεί όταν το Βιετνάμ δεν ακολουθεί τι δεσμεύσει του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα λόγο στα υπόλοιπα μέλη τη ε, επιτροπή Η κυρία Κατάιναν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά σημαντικό το θέμα που εξετάζουμε. Σίγουρα τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελέσουν ένα βασικό σκέλος της ε, συμφωνίας αυτής ελεύθερων συναλλαγών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να γίνουν πρόσχημα για να παρακολύσουμε την έγκριση της συμφωνίας. Φυσικά πρέπει να τηρούνται ε, οι κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμως και ο Επίτροπος Χόργαν, τον οποίο ακούσαμε χθε, ανησυχούσε για τα θέματα προστατευτισμού Πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε πώς μπορούμε να τον ε, αντιμετωπίσουμε. Φυσικά θα είναι καλό για τι εταιρείε μα. Η συμφωνία αυτή θα φέρει περισσότερε θέσει εργασία, αλλά και η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πλέον σημαντική. Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή τώρα. τι θέλουμε τη συμφωνία αυτή και να βοηθήσουμε το Βιετνάμ να προχωρήσει ή θα αφήσουμε την Κίνα να το υποκαταστήσει και να αναλάβει τα, το πρωταγωνιστικό ρόλο. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ως μέλος της αντιπροσωπείας ΑΖΕΑΝ στην προηγούμενη θητεία και επειδή είμαι εξοικειωμένος με αυτή την περιοχή, και ως εισηγητής για τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη που κράτησε πολύ καιρό μέχρι να φτάσουμε σε ακύρωση, παρόλα αυτά την είχαμε δει ως μια, μια πύλη για να έχουμε πρόσβαση, την υψηλή πύλη για να έχουμε πρόσβαση στις χώρες ΑΖΕΑΝ, τώρα έχουμε τη δεύτερη περίπτωση για αυτή τη γεωγραφική περιοχή του κόσμου. Όπως το είπε και η συνάδελφος, το Βιετνάμ και άλλες χώρες ΑΖΕΑΝ θέλουμε να είναι οικονομικός και κοινωνικός ισχυρές για να είναι και ένα αντιπελωδέως για την Κίνα. Ένα ανάχωμα για την Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν να τις προωθήσουμε τις συμφωνίες αυτές. Όπως είπαν και άλλοι, ε, είναι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αρκετά σημαντικό. Αλλά έχουμε επίσκεψη σε λίγε εβδομάδε στη χώρα. Εγώ ήμουν στην προηγούμενη επίσκεψη στο Βιετνάμ πριν από λίγα χρόνια και είχαμε συζητήσει με υπουργού ε, όσοι ήταν υψηλόβαθμοι και έπρεπε να συναντήσουμε εκεί, είχαμε ευκαιρίες να θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα και να δούμε γιατί έχει υποβαθμιστεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είπαμε ότι αδειμονούμε να έχουμε μια συμφωνία μαζί τους, αλλά πρέπει να επιληθούν τα θέματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Και είχαμε τότε ήδη θέματα με τις επιδόσεις τους στην προστασία των δικαιωμάτων. Μα είχαν υποσχεθεί να βελτιώσουν την κατάσταση. Ο Επίτροπο Χόλγκαν πιστεύω ότι μπορεί να το προωθήσει ε, περαιτέρω εφόσον συναυθεί η συμφωνία. Νομίζω θα είναι επιζήμιο για την εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάπτουμε συμφωνίε και μετά να μα παίρνει χρόνια επί χρόνων να τι κυρώσουμε. Όπω έγινε τελικά με τη Σιγκαπούρη. Ευχαριστούμε πολύ. Η Μακουλάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που ανέφεραν όλοι, υπάρχει ανησυχία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε αυτά που είπε η κυρία Γιόρντ Ντάρλινγκ, ε, η σκιώδη συγκίτρια, ότι είχε αυξηθεί από το 2012 και μετά ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων μας. Το 2017 η κυρία Μάλστρομ έστειλε μια επιστολή ε, στην ομόλογό της στο Βιετνάμ ε, με κάποιες ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Ποια ήταν η συνέχεια, πώς θα μπορούσαμε τελικά να εφαρμόσουμε αυτά που αναφέρονται στη συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα την εργασιακή κατάσταση, είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί μια συμφωνία που να επιτρέπει την ελευθερία δημιουργίας ενώσεων και ε, να, να γίνουν αυτά τα εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχουν ανεξάρτητα συνδικάτα. Πώς βλέπετε τα πράγματα για το θέμα αυτό με το Βιετνάμ και με βάση ποιο χρονοδιαγράμμα θα, θα μπορέσει το Βιετνάμ να έχει πραγματικά συνδικάτα. Η νέα ε, εργασιακή νομοθεσία επίσης του Βιετνάμ ε, τι χρονοδιάγραμμα έχει, πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμη πριν τη σύναψη της συμφωνίας. και ο κύριος Βίνκλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, αξιότιμη συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίω για την παρουσίαση και όλε τι πληροφορίε που μα έδωσε. Κάποια θέματα εμπορικά τέθηκαν, όχι τόσα, αλλά να προσθέσω κι εγώ ένα. Αν κατάλαβα καλά, υπάρχει μια εμπορική επιτροπή ε, για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθερών Συναλλαγών που θα θεσπιστεί ε, γνωρίζετε ότι το κοινοβούλιο αυτό να είναι όλο και, θέλει να είναι όλο και πιο ενεργό κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής. Στην επόμενη λοιπόν ε, θητεία του Κοινοβουλίου αλλά και της Κομισιόν στην DigiTrade όλοι θα είναι πολύ προσεκτικοί διότι η παρακολούθηση και οι αρμοδιότητες μας επί παρακολούθηση θα τις ασκήσουμε. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της εφαρμογής διότι η εφαρμογή είναι το σημείο κλειδί. Χωρίς εφαρμογή δεν γίνεται τίποτα. Ούτε οι εμπορικοί στόχοι μας επιτυχάνονται, ούτε οι, άλλοι στόχοι μας. Νομίζω αυτή η Επιτροπή θα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο και θα δημιουργηθούν κάποιες ομάδες εργασίας, εργασίες και κάποιες ειδικέ επιτροπές ε, σε επιμέρους τομείς, σε ζητήματα πρόσβαση στην αγορά, στην αγορά που είναι πολύ σημαντικό για τις δικές μας ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ε, οι εταιρείε ε, είναι άλλωστε ο πιο σημαντικό εταίρο μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και βεβαίω υπάρχει και η ρυθμιστική συνεργασία που είναι σημαντική. Ε, Πώ λοιπόν αυτή η επιτροπή θα δίνει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, ποια θα είναι δική μας, ο δικό μα σύνδεσμο με αυτήν την επιτροπή. Θα έρχονται εδώ στο Κοινοβούλιο, θα ενημερωνόμαστε για την εφαρμογή ή εσεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας δίνετε αναφορά στο όνομα της Επιτροπής αυτής εκ των Ευχαριστώ πολύ. Πολλά ε, και διάφορα είπαν οι συνάδελφοι. Πολλές απαιτήσει από τη βιετναμική πλευρά ε, σε ό,τι αφορά ανθρώπινα δικαιώματα, τις συμβάσεις ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας, ε, εμείς ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να, ακολουθηθούν, να ακολουθεί ο σωστός δρόμος. Δεν υπάρχει χρονική πίεση, θα συζητήσουμε τη διαδικασία ε, και απευθύνομαι στην, στην, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω ε, να επαναλάβω το ο κ. Βίνκλερ. το Δημοκρατικό Όργανο του Ευρωπαϊκού πρέπει να μπορεί να εποπτεύει αυτές τις εφαρμογές. Υπάρχουν ε, πολλές συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών με κοινέ επιτροπές που είναι εντελώς απομονωμένες από τον πραγματικό κόσμο. Ε, χρειαζόμαστε δημοκρατική διαφάνεια ε, κατά τη διαδικασία υλοποίηση, κατά τη διαδικασία εφαρμογής. Και θέλουμε πραγματικά να ξέρουμε πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ, Μπέρντ. Και ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων, έτσι να πιάσω λίγο και τον παλμό ε, των μελών της Επιτροπής αυτής, πέρα βεβαίως από την οικονομική σημασία της συμφωνίας, εδώ όλοι συμφωνούμε, Προφανώς ε, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα ε, στα πιο τομεακά ζητήματα, γεωγραφικές ενδείξεις. Εδώ έχουμε την προστασία 196 ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων μέσω της συμφωνίας αυτής. 169, 169 γεωγραφικές ενδείξεις ευρωπαϊκές που προστατεύονται. Αποτελούν μέρος της συμφωνίας, προστατεύονται από τη συμφωνία σε επίπεδο προστασίας ε, συγκρίσιμο με αυτό που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τη Σιγκαπούρη ήταν πιο δύσκολη διαδικασία αυτή, εδώ οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύονται μέσω της συμφωνίας αυτής. Για τους ενδεχόμενους κινδύνους ε, ε, ότι δηλαδή θα μπορούσε αυτή η συμφωνία να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να δοθεί προτίμηση σε προϊόντα που δεν προέρχονται από το Βιετνάμ. Εδώ έχουμε ένα πρωτόκολλο προέλευσης πολύ λεπτομερές, 200 σελίδων, που ε, εξηγεί πολύ, πολύ λεπτομερώς τι σημαίνει ένα προϊόν βιετναμέζικης προ... Ε, προέλευσης και ένα προϊόν ευρωπαϊκής προέλευσης. Για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν παρατυπίες, υπάρχουν διατάξεις πολύ συγκεκριμένες για τους αγωγείς, τους εξαγωγείς, αλλά και διοικητική συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών, τελωνιακών αρχών, για να αντιμετωπιστούν οποιασδήποτε παρατυπίες στο ζήτημα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα το IUU και την αλία ήμουν στην Επιτροπή Αλίας και εκεί είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Στην Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών υπάρχει ένα άρθρο εξαιρετικά ισχυρό, το άρθρο 38, ε, για τα ζητήματα ακριβώ της αλίας, της βιώσιμης αλίας, που αναφέρεται σε συνεργασία για να αντιμετωπιστεί η αλία IUU, η παράνομη αλία δηλαδή, ε, και να, για να εξασφαλίσουμε μια σωστή διακυβέρνηση στον τομέα της αλίας παγκοσμίω εφαρμόζοντας ε, τις αρχές που διέπουν τις διεθνείς συμφωνίες. Η δέσμευση αυτή στον τομέα της αλίας ε, θα ενισχύσει την ε, συμφωνία που υπάρχει για την αλία IUU με το Βιετνάμ. Υπάρχει κίτρινη κάρτα βέβαια προ το Βιετνάμ ως χώρα που δεν συνεργάζεται στην καταπολέμηση αυτή της μορφής Αλίας. Βεβαίω είναι μια άλλη διαδικασία αυτή. Ε, οι συμπληρωματικέ μεταξύ του δύο διαδικασίε αναμένουμε τα αποτελέσματα της πίεσης που ασκείται στο Βιετνάμ από τους συνάδελφους ε, της DG Mario στα πλαίσια της, ε, του κανονισμού IUU ε, τον Νοέμβριο. Τώρα για τα εργασιακά. Ε, ανεξάρτητα συνδικάτα. Με βάση τον εργασιακό κώδικα που ελπίζω να μας τον φέρετε όταν θα επανέλθετε ε, αναγνωρίζονται τα ε, ε, ανεξάρτητα συνδικάτα. Επίσης το Βιετνάμ έχει δεσμευτεί ως το 2023 να επικυρώσει την ε, σύμβαση του 87 για τις ανεξάρτητα συνδικάτα. Ναι, τώρα, τώρα έρχομαι στην εφαρμογή, στο θέμα της εφαρμογής. πρώτα όμως να μιλήσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλοί επικεντρώθηκαν στο θέμα αυτό και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε απολύτως την κατάσταση στο Βιετνάμ. Δηλαδή ελπίζω να αντιλαμβανόμαστε απολύτως την κατάσταση. Ε, και ε, προφανώς είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο εσά, αλλά και εμά, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε κατά νου από πού έρχεται αυτή η χώρα. Και έχει σημειωθεί πρόοδο ε, ιδίω στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα. Εμεί ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο τη εμπορική μα πολιτική. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσει απέναντι στο Βιετνάμ. Αυτό είναι μια βασική αρχή ε, στι σχέσει μα με το Βιετνάμ εδώ και δεκαετίε. Υπάρχει άμεση νομική διασύνδεση ε, δεσμευτική ε, μεταξύ της Συμφωνίας των Τέρων και και τη Συμφωνία ε, σύμπραξης. Εάν λοιπόν υπάρξει παραβίαση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, ε, μπορούν και οι δύο αυτές συμφωνίες να προσβληθούν. Υπάρχει συνεργασία στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του διαλόγου για ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε σε βάθος συνταλλαγέ απόψεων και έχουμε και άλλη μια ευκαιρία να προωθήσουμε ε, τις, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των δημοσίων δηλώσεών μας έγινε αναφορά στην επιστολή τη κυρία Μάλμστρομ Ερχόμαστε σε επαφή με υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχει συνεργασία στο τομέα τη ανάπτυξη και σχετικά project και το ευρωπαϊκό project, ευρωπαϊκό όργανο μάλλον για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών εκεί και να προστατεύσουμε τι ευάλωτε ομάδε. Έχουμε ειλικρινή συζητήσει με το Βιετνάμ και για το θέμα τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η εφαρμογή του FTA θα μας δώσει περαιτέρω εργαλεία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το διάλογό μας με το Βιετνάμ και να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος ε, για τα εργασιακά δικαιώματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερο κράτος δικαίου και μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη δημιουργία νέων διάβλων, διάβλων επικοινωνίας με τις αρχές του Βιετνάμ. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, Πρόεδρε, Βεβαίω παραδοσιακά υπάρχει μια δομή εφαρμογή στα πλαίσια ε, τη τηλεφωνία των Συναλλαγών, η οποία ενεργοποιείται αφού υπογραφεί η συμφωνία. Υπάρχουν και εξειδικευμένε επιτροπέ που παρακολουθούν την ε, εφαρμογή και από τι δύο πλευρέ. Ε, στην περίπτωση προβλημάτων ε, υπάρχει και διαδικασία επίλυση διαφορών. Θα υπάρχει ένας επικεφαλής για την εφαρμογή. Ε, θα τον επιλέξει ο νέο επίτροπος, ο κ. Χόγκαν αναμένουμε να δούμε πώς θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την αναφορά που θα πρέπει να δώσουμε για τα αποτελέσματα των συζητήσεων στα πλαίσια των διαφόρων επιτροπών FTA και με βάση και τον επικεφαλής δηλαδή για την εφαρμογή. Μια και είναι εδώ η συνάδελφος η Μαντέν Τένιγκερ που παρακολουθεί τα ζητήματα εμπορίου και βιώσιμη ανάπτυξη έχει και αυτή δύο λόγια να πει για την πτυχή της τεχνικής συνδρομής και την εφαρμοστικότητα αυτού του κεφαλαίου. Ευχαριστώ, Πίτερ. Καλημέρα. Υπογράμμισες ε, τα βασικά πολύ ωραία. Να πω κι εγώ κάτι. Ένα παράδειγμα από τα προηγούμενα χρόνια που μου ήρθε ακούγοντάς ε, ε είχαμε μια πολύ καλή αποστολή το 2017 που είσαστε και εσείς κύριε Λάγκε και όταν πήγαμε δεν υπήρχε τίποτε. Υπήρχαν κάποια μηνύματα ενθαρρυντικά, αλλά πρακτικά τίποτε. Αυτό που έγινε μέσα σε δύο χρόνια είναι πάρα πολύ ισχυρή μόχλευση. Εμείς το παρακολουθήσαμε. Θα πάμε και μετά από εσά το Νοέμβριο. Ε, μιλάμε ήδη για την δημιουργία του TST Board, για την κοινωνία των πολιτών, μιλάμε για εκπαίδευση, μιλάμε για προτεραιότητες, κλίμα, θέλουν να δουλέψουν μαζί μας για το κλίμα. Υπάρχουν πολλά στον τομέα των εργασιακών. Είχαμε μεγάλες διαμάχες και με το ILO, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, και επίσης χρειάζονται και τεχνική ε, βοήθεια. Είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να αναλάβουμε δέσμευση για να αναλάβουν μετά και αυτοί. Το η που επεξεργαζόμαστε με την ε, ILO ε, αφορά το Βιετνάμ. Μιλάμε για ενέργειες που θα ενδυναμώσουν πολύ τις προσπάθειές μας σε αυτούς τους τομείς. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι ε, πρέπει να δούμε εκεί που πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Και θα το δείτε και επί τόπου όταν πάτε για την ελευθερία του συνέρχεσθε. Ε, ε, εκεί ε, θέλουν, θέλουν ελευθερίες, θέλουν να μπορούν να συνέρχονται ειρηνικά. Αυτό το δήλωσαν, ανέλαβαν δέσμευση και θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας για να τα επιτύχουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν η πρόσκληση αυτή πρέπει να βρει ανταπόκριση από μας ώστε να ισχύσουν αυτά στην πράξη. Ε, είναι ένα από τα σημαντικά η ελευθερία του συνέρχεστε. Τώρα για την επιβολή παρακολούθηση και επιβολή, ε, αυτό είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Πρέπει να τα, τους παρακολουθούμε όλους. Υπάρχει ε, αναφορά στην ε, συμφωνία. δεν αφορά μόνο την Κομισιόν, αλλά και επιτόπου την παρακολούθηση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους μοχλούς που έχουμε ο, υπάρχει επικεφαλής ε, υπεύθυνος ε, για την παρακολούθηση και την ε, επιβολή των μέτρων. Θα προσδιοριστεί η εντολή του ή της, ανάλογα ποιος θα είναι. Τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο, όταν πήγαμε το Μάιο, μιλούσαν για την επίσκεψη του κυρίου Λάνε, Είναι σημαντικό να ε, υπάρχουν αποστολές από το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό γιατί περνάει το μήνυμα ότι τους βοηθάμε και βοηθάτε και μας. Ε, επίσης, ε, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η ιδέουσα επιμέλεια, όλα αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν και είναι αντικείμενα συζήτησης μεταξύ επιχειρηματιών Ευρωπαίων και Βιετναμέζων. Ε, επίσης πρέπει ε, και με την ε, επεκτείνεται θέματα με δέουσας επιμέλειας, τους απασχολούν και λένε ότι πρέπει να τα συζητήσουν και με την Κίνα, γιατί δεν είναι υπεύθυνοι για το τι κάνουν εκείνοι. και άλλοι εταίροι, είπα, ο Καναδάς, ενεργοποιούνται και συνεργάζονται και εκείνοι για όλα αυτά τα θέματα με το Βιετνάμ. Ε, πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προετοιμάσουμε το Βιετνάμ για να μπορεί να προχωρήσει σε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση που θέλουν να κάνουν σε εργασιακά και άλλα θέματα. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση ε, συμπληρωματική από την Ίνα Ροντρίγκες. Ναι, είναι αλήθεια ότι το Βιετνάμ έχει κάνει σημαντικά βήματα, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι μένουν πολλά να γίνουν. Ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι όταν έχουμε συστηματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούσε να υπάρξει ε, αναστολή της προτιμησιακής πρόσβαση στην αγορά. Τι εννοείται συστηματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποιο το ορίζει αυτό. Και όταν διαπιστωθεί, διαπιστωθεί αυτό, τι ακριβώς θα γίνει και τι ρόλο θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο καθορισμό ε, της διαπίστωσης αυτής ε, της παραβίασης. Ε, κυρία Τσάουνς. Ευχαριστώ. Συνεχίζω πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που θέλω με πρόοδο πριν κυρώσουμε όχι υποσχέσεις τι θα γίνει το 2023. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις, πολιτικοί κρατούμενοι, μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα κλπ. Ένα άλλο θέμα είναι η παιδική εργασία. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, περίπου 10% των παιδιών στο Βιετνάμ δουλεύουν και ένα τρίτο δουλεύει full time. Ε, έχουμε τα στοιχεία και ο αρμόδιος επίτροπος είπε ότι θα δείξουμε μηδενική ανοχή σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα θέμα όπου πρέπει να έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο πριν προχωρήσουμε στην συμφωνία. Να μιλήσω πρώτα για την παιδική εργασία. Ναι. Ναι, και αυτό συζητείται πλήρως θα δείτε στην αποστολή που θα πάει στο Βιετνάμ, θα δείτε ότι αυτό το έχουμε ε, ως προτεραιότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, αφορά την οικονομική κοινωνική δομή. Η Κομισιόν εργάζεται επί ενός προγράμματος δράσης που θα είναι έτοιμος το Δεκέμβριο. Το συζητούμε μαζί τους σε πλήρη συνεργασία με την ILO. Κοιτάζουμε λοιπόν το θέμα για να δούμε πώς θα τους βοηθήσουμε. Υπάρχει και σύσταση από την ILO σχετικά με την παιδική εργασία. Οπότε εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί πλήρως η σύμβαση του ILO που αφορά την παιδική εργασία και την απαγορεύει. Η παιδική εργασία είναι κάτι διαφορετικό από την ελευθερία του συνέρχεστε και θα πρέπει να ε, συζητηθεί χωριστά. Υπάρχουν ε, στοιχεία που μπορώ να σας στείλω. Ε, σίγουρα το θέμα είναι μεγάλη προτεραιότητα. Η παιδική εργασία για μας είναι πολύ υψηλή προτεραιότητα και το παρακολουθούμε και το συζητούμε και ε, τώρα συντάσσουμε και ένα πρόγραμμα δράσης, σχέδιο δράσης. Ναι, να συμπληρώσω κάτι. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που αναστέλουν τις ε, παραχωρήσεις ε, σε μια συμφωνία ή και αναστολή όλης της συμφωνίας. Αλλά ε, το, εμείς μιλάμε για κατάλληλα μέτρα. Αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί και με τα άλλα θεσμικά όργανα για να δούμε ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα. Η αναστολή θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση, η, η, η ίστατη καταφυγή αλλά βέβαια η απειλή υπάρχει ότι δηλαδή εάν υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις κατά χρήσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων τότε ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ. Ευχαριστώ. Και ο αντικαταστάτης εισηγητής μας, μήπως θέλει ε, να προσθέσει κάτι κύριε Φράγκο, ναι. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος τους Γιάν. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις σε αυτό το στάδιο. Θέλουμε καταρχήν να ρωτήσουμε τι πληροφορίες έχει συλλέξει η Κομισιόν από τα κράτη-μέλη σχετικά με την έγκριση της συμφωνίας. Ε, εδώ πρόκειται για το κλείσιμο της πρώτης συζήτησης. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις άλλες σε αυτό το στάδιο, κλείνουμε το εμπορικό κομμάτι, αν θέλετε. Ε, Πίτερ, νομίζω δεν απαντήθηκε η ερώτηση του κυρίου Βίνκλερ. Καλά. Ε, ε, θα, θα μας ενημερώσετε κάποια στιγμή αργότερα για να μπορεί να συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία και το Κοινοβούλιο. Εγώ προσβλέπω στη ε, καθοδήγησή σας. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι αφορά τις επενδύσεις. Και ο εισηγητής τώρα θα μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή. Έχουμε μισή ώρα για αυτό το θέμα. Και δίνω το λόγο στον κύριο Φράγκο. Τώρα είναι το δεύτερο κομμάτι και η ερώτηση. Ε, ήθελα να ρωτήσω τι πληροφορίες έχουν, έχει συλλέξει η Κομισιόν από τα κράτη-μέλη σχετικά με την έγκριση της Συμφωνίας Επένδυσης από τα Εθνικά Κοινοβούλια και αν ήρθε σε επαφή η Κομισιόν ε, αν γνωρίζει πόσο θα αυξηθούν οι επενδύσεις στο Βιετνάμ και ποιες είναι οι μεγάλες δυσκολίες που αναφέρονται από τις επιχειρήσεις μας. Με συγχωρείτε που... Μάλιστα, σύντομα μας τα είπατε. Και τώρα δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Η Μαρία Μάρ... Μάρτιν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω μια ανασκόπηση σύντομα της ε, Συμφωνίας Προστασίας των Επενδύσεων και αν θέλετε μετά θα απαντήσω και στις ερωτήσεις του εισηγητή. Σχετικά με τη Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων είναι δεύτερη φορά που ερχόμαστε σε αυτή την Επιτροπή με μια τέτοια συμφωνία που ακολουθεί τη νέα αρχιτεκτονική που εφαρμόζουμε για πρώτη φορά με τη Σιγκαπούρη και σας ενημερώσαμε την τελευταία φορά. Εδώ συζητούμε για μια συμφωνία που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών, της ΣΕΣ. Και ακολουθεί τη θεσμική και πολιτική δομή η οποία ε, θεσπίζεται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Αυτά είναι βασικά για τις επενδύσεις. Στη Συμφωνία ΣΕΣ ε, θέλουμε πρόσβαση στην αγορά γιατί διασφαλίζομαι, απελευθέρωση του ε, εμπορίου και επίσης ε, επίπεδο προστασίας των επενδύσεων, στη Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων και επίλυση διαφορών. Και οι δύο συμφωνίες είναι φιλόδοξες από την άποψη των επενδύσεων. Είναι σημαντικός αυτός ο προορισμός για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και δεν θα έπρεπε να ε, δίνουν προνομιακή θέση στους επενδυτές μας, αλλά να εξασφαλίζουν ίσους όρους του παιχνιδιού στις ε, λειτουργίες με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα και συνθήκες αγοράς που δεν δημιουργούν διακρίσεις και είναι δικές. Είναι σημαντικό και γνωρίζω ότι αυτό είναι βασικό για σας και πρέπει να το επαναλάβουμε άλλη μια φορά, ότι η Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων και η προστασία που χορηγείται μέσα από αυτή τη συμφωνία διασφαλίζει το δικαίωμα ε, ρύθμισης των μερών και να ε, ε, προωθούν στόχους θεμητούς Επίσης είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε την μεταρρύθμιση, εξυγχρονισμό του συστήματος επενδύσεων και να υπάρχει και κατάλληλο σύστημα επίλυσης διαφορών. Ε, το έχουμε ξανασυζητήσει στο Κοινοβούλιο αυτό το θέμα. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα κέριο στοιχείο της συμφωνίας που θα μας βοηθάει να αντικαταστήσουμε 21, 21 21 συμφωνίες σε διμερές επίπεδο μεταξύ χωρών και να έχουμε ένα σύστημα ε, επίλυσης διαφορών για όλους. Θα υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα για τις επενδύσεις που θα προωθεί την διαφάνεια, την αμεροληψία και θα ε, προσφέρει και εγγυήσεις. Επίσης ε, παρέχει όλα τα στοιχεία που επιβεβαίωσε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι είναι απαραίτητα για τέτοιου είδους συμφωνίες, γιατί γνωρίζετε την απόφαση για την συμφωνία ΣΕΤΑ που δεν είχε ληφθεί από το δικαστήριο όταν συζητούσαμε τη Σιγκαπούρη. Τώρα όμως ε, έχουμε την απόφαση με όλες τις συνιστώσεις της και μπορούμε να τη λάβουμε, και θα τη λάβουμε υπόψη μας ε, για να αντιμετωπίσουμε τυχόν διαφορές και αποκλήσεις από τον νόμο της το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων θα πρέπει να έχει τα ίδια, τις ίδιες αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως υπάρχουν και στην ΣΕΣ ε, και αναφέρθηκαν στην εισαγωγή μας ε, νομοθετικό πλαίσιο ε, που θα προβλέπει όλα αυτά. Τέλος, να υπογραμμίσω τη συμφωνία αυτής της συμφωνίας όχι μόνο ως κομμάτι της ε, συμφωνίας για το εμπόριο ε, που θέλουμε να έχουμε με το Βιετνάμ, αλλά και ως ένα βήμα ε, εφαρμογής της προστασίας των επενδύσεων και επίλυσης των διαφορών. Είναι σημαντικό να έχουμε μία ακόμα δικαιοδοσία στο πλευρό μας για να αντιμετωπίζουμε θέματα ε, των επενδύσεων. Ε, ελπίζω να προχωρήσει η διαδικασία κύρωσης. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω, θέλετε να απαντήσω και στις ερωτήσεις ε, που τέθηκαν ε, από τον εισηγητή. Ναι, αργότερα. Μισό λεπτό να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι σκιώδεις έχουν το λόγο. Ο κύριος Χάνσεν αντικαθιστά τον σκιώδη του ΕΛΚ. Δεν θέλω να κρατήσει πάρα πολύ άλλο η συνεδρίαση. Η παρουσίαση ήταν διεξοδική, οπότε θα αφήσω τις ερωτήσεις στον εισηγητή. Δεν είμαι εγώ ο υπερκεφαλής και όδης από την ομάδα μου. Ας ε, θέσει τις ερωτήσεις του ίδιου ο εισηγητής. Ευχαριστούμε κυρία Κεταντάλη. Και εγώ συνοπτικά. Πολλές από τις ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών αφορούν και αυτά για, για τις επενδύσεις, η οποία επικεντρώνεται στα δικαιώματα των επενδυτών κυρίως και πολύ λιγότερα έχει για τις υποχρεώσεις των επενδυτών. Η Μάτλιν είπε στη συζήτηση για το TST τη δέουσα επιμέλεια Και εδώ ε, μας ενδιαφέρει αν μπορείτε να μας πείτε τίποτα λεπτομέρειες για την επενδυτική συμφωνία και πώς αυτό διασυνδέεται με την δουλειά που γίνεται για το TST. Για τις επενδυτικές λοιπόν σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ βλέπετε να υπάρχει ε, μεγάλη ροή άμεσων επενδύσεων, απευθείας επενδύσεων ε, προς τις, χώρες, τις τρίτες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τεμερείς συμφωνίες. Από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κάριν δεν είναι εδώ. Για τους πράσινους η κυρία Σφόντ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ γρήγορα για το θέμα για τη συμφωνία αυτή των επενδύσεων. Τι διατάξεις περιέχει σε περίπτωση που το Βιετνάμ βελτιώσει εντωμεταξύ τις κοινωνικές του και περιβαλλοντικές του προδιαγραφές. Μήπως τιμωρηθεί βάσει των προηγούμενων διατάξεων η χώρα αυτή. Πραγματικά εκπλήσω με πολύ σύντομες ερωτήσεις. και ο κύριος Λατσίνη. Κύριε Λατσίνη, δεν είχα ζητήσει το λόγο, αλλά θα υποφεληθώ. Είχαμε, έχουμε τα ίδια προβλήματα, πιστεύω, που είχαμε και προηγουμένως. Μια σειρά από θετικές προτάσεις που όμως δεν ε, συνοδεύονται από υποχρεώσει. Δηλαδή δικαιώματα ωραία αναφέρονται, αλλά δεν υπάρχει πουθενά η αναφορά στην υποχρέωση σεβασμού των δικαιώματων αυτών και πώ τα παρακολουθείτε. Ευχαριστούμε κύριο Σόλτ. Είμαι βέβαιο ότι θα εξαντλήσει το δίλεπτο. Σου δίνω ένα επιπλέον λεπτό. Ένα λεπτό μόνο, μα ήταν αρχικά δύο τα λεπτά. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και σχολιάζοντα τα ερωτήματα των σοσιαλιστών και πρασίνων. Η ιστορία της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του Βιετνάμ είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς θα βεβαιωθείτε ότι θα έχουμε ισότιμες σχέσεις και δίκαιο ανταγωνισμό στις, ε, στους επενδυτές που θα λειτουργούν στο Βιετνάμ. Πρέπει να κοιτάμε και προς το μέλλον δεν είναι το πρόβλημα αν θα έχουμε ε, μηχανισμό διατησία ή μηχανισμό διαμεσολάβηση του ενό του άλλου τρόπου. Ε, το θέμα είναι να είναι επενδυτέ ε, πιστοί στι υποχρεώσει του. Επίσης, θέλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και υπερβολοντικά πρότυπα να είναι κάτι που θα υπερτερεί τον δικαιώματα των διτών είτε σε αυτή τη συμφωνία είτε μέσω των ρητρών των διεθνών συνθήκων όπως αυτή που διαπραγματεύεται η διακυβερνητική ομάδα για τα δικαιώματα αυτά στην Γενέβη, στον ΟΗΕ. Να έχουν δικαιώματα δηλαδή οι επενδυτέ, δεν λέμε, αλλά να έχουν και υποχρεώσει για να είμαστε βέβαιοι ότι προστατεύονται οι πολίτε τη εκάστοτε χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριο Βίνκλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω χρόνο να κάνω και ένα σχόλιο και μετά μια ερώτηση. Διότι το σχόλιο μου αφορά και πάλι το θέμα της προστασίας των επενδυτών. Να θυμίσω στους αγαπημένους συναδέλφους μου ότι παρά τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, πολλά προβλήματα δεν έχουν επιληθεί. Η χώρα που, έχω, γνωρίζω εγώ πολύ καλά, συνήθως βρίσκεται στην αδύναμη πλευρά των διμερών αυτών σχέσεων, των συνθήκων αυτών. Και το λέω μόνο και μόνο για να είναι ξεκάθαρο. Ε, Επιτροπή, πολύ σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίε αυτές για, για την επενδυτική συμφωνία σε συνεργασία με το Βιετνάμ. Θα ήθελα να θέσω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Η Επιτροπή μας θα πάει επίσκεψη στο Βιετνάμ, όπως ξέρετε, σε λίγες εβδομάδες. Θα είμαστε εκεί. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το βασικότερο μήνυμα που πρέπει να περάσουμε εκεί στους πολιτικούς ευθύνοντες διότι είναι χώρα σοσιαλιστική. Αλλά μας ενδιαφέρει να απευθυνθούμε σε όλους τους ενδιαφερομένους, να έχουμε επαφή με όλους τους συνομιλητές και κυρίως να αγγίξουμε τους πολιτικούς ηθήνοντες που αυτή τη στιγμή έχουν την εξουσία. Ποιο θα ήταν το δικό σας πολιτικό μήνυμα, τι πιστεύετε ότι να περάσουμε. Ευχαριστούμε και τώρα η σειρά σας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να τις ομαδοποιήσω για να απαντήσω εντός του χρόνου που μας έχει μείνει. Ε, για το βασικότερο σημείο που έχετε θίξει πολλές ερωτήσεις για την επενδυτική συμφωνία αυτή, καθή, αυτή και το πώς επιτρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι τι πλαίσιο προβλέπουμε εδώ για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Όπως σας είπα, η πρόσβαση στις αγορές καλύπτεται ούτως ή άλλως και από τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Πρέπει λοιπόν να τα συνδυάσουμε τα δύο, να τα δούμε παράλληλα. Στην Συμφωνία των Επενδύσεων δηλαδή μετά. Είναι πιο σημαντικό για τη συζήτηση που κάνουμε ότι οι επενδύσεις ουσιαστικά δεν διαφεύγουν από μια χώρα. Τις διατηρούν. Δηλαδή λόγω των ε, υποχρεώσεων πρόσβαση στις αγορές που προκύπτουν από τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών μπορεί να γίνει πιο ελκυστική αγορά μιας χώρας, όμως χάρη στην επενδυτική συμφωνία γίνεται σταθερό το περιβάλλον, γίνεται ευνοϊκό δίκαιο, δίκαιος προς τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες, αυτό βοηθάει. Οι επενδυτές μένουν. Και έτσι υποφελείται όχι μόνο η χώρα της επένδυσης, αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το ρόλο των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κυρώσουν την ε, Συμφωνία για την Προστασία των Επενδύσεων. Είναι μια μεικτή συμφωνία και μόλις δώσετε τη συγκατάθεσή σας θα αρχίσουμε τη διαδικασία κύρωσης από όλους, ε, όλους τα αρμόδια εθνικά κοινοβούλια. Και βεβαίως αυτή είναι μια διαδικασία, όπως πολύ καλά γνωρίζει αυτός ο οίκος, παίρνει χρόνο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κυρώσεις, αν κατάλαβα καλά το ερώτημα, έτσι, οι αρνητικές επιπτώσεις για τα επίπεδα προστασίας, παραδείγματος χάρη, ε, σε περιβαλλοντικό επίπεδο, σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λόγω της προστασίας ε, επενδύσεων και της σχετικής συμφωνίας, εμείς δεν θεωρούμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, προσέχουμε και φροντίζουμε να έχουμε πολύ σαφείς διατάξεις για το δικαίωμα ρύθμισης. Έχουμε διατάξεις που προβλέπουν ότι τα συμβολόμενα μέρη δεν μπορούν να κατεβάσουν τον πύχη της προστασίας για να προσελκύσουν επενδύσεις και βεβαίως είμαστε πεπισμένοι ότι το FDI και το API από κοινού μπορούν να βοηθήσουν για να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις που λαμβάνουν χώρα στο Βιετνάμ συμμορφώνονται με το ε, απαιτούμενο επίπεδο προστασίας ε, σε περιβαλλοντικό επίπεδο, σε εργασιακό επίπεδο, σε επίπεδο εταιρική ευθύνη και ότι το Βιετνάμ, όπως ελέγχθη νωρίτερα, θα κάνει τις απαραίτητες ε, νομοθετικές αλλαγές σε επενδύσεις ε, που θα γίνει στο έδαφος του θα γίνουν επί της σωστής βάσης. Να σας θυμίσω εν συντομία ότι στο IPA δεν επαναλαμβάνουμε απλώς τις, ε, την θεμελιώδη, τη Σύμβαση Θεμελιώδη Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση των Εθνών. Μιλάμε και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μιλάμε και για τη διαφάνεια. Όλα όσα δηλαδή περιλαμβάνονται και στο FTA. Επίσης και αυτό είναι σημαντικό, το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, καθιστούμε σαφές ότι προστατεύουμε τους επενδυτές οι οποίοι συμμορφώνονται με την εσωτερική νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε το επίπεδο εσωτερικής ρύθμισης. Θέλουμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία του Βιετνάμ για τις υπεύθυνε επενδύσεις. Ταυτόχρονα λέμε ότι θα προστατεύσουμε μόνο τους επενδυτές εκείνους οι οποίοι ε, δρούν υπεύθυνα και συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Δεν προστατεύουμε επενδυτές που δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία του Βιετνάμ. Αυτήν δηλαδή προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Επίσης είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι τα συμβαλόμενα μέρη θα αναλάβουν δεσμεύσεις για να προωθήσουν στο FDA και στο API ε, για υπεύθυνε ε, συμπεριφορές των επιχειρήσεων αυτή είναι μια δουλειά που γίνεται και στο επίπεδο εφαρμογής. Ήδη σε αυτή τη φάση υπάρχει ένα project για μια υπεύθυνη αλυσίδα εφοδιασμού. Δεν ξέρω αν ξέχασα τίποτα, Πρόεδρε. Θα μου το θυμίσετε, αν έχω ξεχάσει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι ακόμα. το μήνυμα και ο κύριος Βίνκλερ, ναι, είχα ξεχάσει πώς ε, το ξέχασα για το μήνυμα. Σε ό,τι αφορά το κεντρικό μήνυμα, πρέπει να επιμείνουμε στην ανάγκη βελτίωσης όπως γίνεται και στα πλαίσια του FTA, την νομοθεσία έτσι ώστε να συμμορφωνόμαστε με τους στόχους του εμπορικούς, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να το συνδέσουμε αυτό με το γεγονός ότι εμείς θέλουμε επενδύσεις στο Βιετνάμ που να συμμορφώνονται με υψηλό επίπεδο προστασίας για τα περιβαλλοντικά και, περιβαλλοντικά εργασιακά ζητήματα. Δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τη συζήτηση μεταξύ του FDA και της Συμφωνίας ε, Προστασίας Επενδύσεων. Το άλλο πολύ σημαντικό μήνυμα είναι η δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε από κοινού για να εφαρμόσουμε ε, το σύστημα επενδύσεων, να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει και βεβαίως ευρύτερα θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία για το σκέλος που αφορά τις πολυμερές επενδύσεις. Τώρα, εάν το Βιετνάμ προχωρήσει, θα έχουμε ήδη τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ με ένα σύστημα επενδύσεων και που θα έχουν συμφανίσει όχι μόνο για τον κώδικα επενδύσεων, αλλά και για τον κώδικα ε, ε, πολυμερών επενδύσεων. Θέλουμε να μπει και ο Καναδάς, θέλουμε να μπει το Μεξικό, θέλουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με την Ιαπωνία. Το βήμα του Βιετνάμ είναι ένα σημαντικό βήμα. Θέλουμε ένα πολιτικό μήνυμα όχι μόνο απέναντι στο Βιετνάμ, αλλά και ευρύτερα προς την περιοχή του Ειρηνικού. Για τα SOEs δεν ξέρω αν θέλουν να πούν κάτι οι συνάδελφοι για το FTA, για το Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών, ένα γενικό σχόλιο, το, τα SOEs, και φαντάζομαι ότι αυτό αφορά τα βιετναμέζικα SOEs, αναμένεται να συμμορφώνονται με την ομοθεσία και το επίπεδο προστασίας που θέλουμε να θεσπίσει το Βιετνάμ. Και αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, η προστασία, ε, η συμφωνία προστασίας επενδύσεων δεν πρόκειται να χορηγηθεί. Είτε μιλάμε για SOEs, είτε μιλάμε για ιδιωτικές εταιρείες. Ε, δεν ξέρω αν θέλει να δώσει το λόγο στον Πίτερ Πρόεδρε, ενδεχομένως θέλει να συμπληρώσει για τις SOEs στο FTA, στη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών. Ναι, ο κ. Σόλτ δεν είναι πια εδώ βέβαια. Α, εδώ είναι. Α, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ακούστε, το FDA δεν λέει στην κάθε χώρα πώς θα οργανώσει την οικονομία της. Πώς θα οργανώσει την κατανομή αρμοδιοτήτων. Ούτε εμείς το δεχόμασταν. Όμως, έχουμε διαπραγματευτεί με το Βιετνάμ ένα πολύ φιλόδοξο κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τι δεσμεύσει για τι SOEs από οποιαδήποτε συμφωνία ελευθερών συναλλαγών. σε ό,τι αφορά τις SOE, κρατικές ε, εταιρείε. Ξέρετε ότι είναι μια πολύ συγκεντρωτική οικονομία η οικονομία του Βιετνάμ. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη συμφωνία αυτή είναι ότι εφόσον υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις οι οποίε δρούν στην αγορά θα πρέπει να ακολουθούν τις ε, εμπορικές, τους εμπορικούς κανόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε ε, ε δεσπόζουσα θέση για να προβούν σε διακρίσει απέναντι σε πελάτε ή άλλου παρόχου. Υπάρχουν διαφα... Ε, διατάξει λοιπόν υπερδιαφάνεια για την ιδιοκτησία, τη δομή και τη συμπεριφορά αυτών των κρατικών οντοτήτων. Αυτά υπάρχουν στη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών. Ευχαριστώ. Δύο ακόμα ερωτήσει. Ο κύριο Κέλλη και ο κύριο Σόλτ. Ευχαριστώ σε σχέση με αυτό που συζητάμε, νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό σύστημα στη Σιγκαπούρη για τη διαφάνεια. Την ανεξαρτησία των συνδικάτων κτλ. Είναι παρεμφερής αυτή η συμφωνία με το Βιετνάμ, με αυτή τη Σιγκαπούρη. Και τα επόμενα πέντε χρόνια, κατά τη της θητείας του κυρίου Χόγκαν, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πολυμερές ε, δικαστήριο το οποίο θα μπορεί να δρά παγκοσμίω. Ο Χέλμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ. Ξαναγυρίζω στο κώδικα για τις επενδύσεις. Πόσο ενεργά συμμετέχει το Βιετνάμ στις διαπραγματεύσεις για την καλύτερη προστασία και προς ποια κατεύθυνση κινείται γιατί μπορεί να είναι δραστήριος εταίρος το Βιετνάμ ε, δημιουργώντας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ πολυμερείς ρυθμίσεις για την προστασία των επενδύσεων. Ευχαριστώ για τις συμπληρωματικές ερωτήσεις σε ό,τι αφορά το αν είναι διαφορετικό το Βιετνάμ από τη Σιγκαπούρη. Όχι, δεν είναι σε σχέση με τις επενδύσεις, ενώ έχει το ίδιο υψηλό επίπεδο διαφάνειας, ανεξαρτησίας που περιέγραψα στην προηγούμενη παρέμβασή μου. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα έχουμε την ίδια μεταχείριση στο Βιετνάμ όπως στη Σιγκαπούρη. Αλλά θα πρέπει να αντικαταστήσουμε 12 ε, ε, επιμέρους συμφωνίες και στη Σιγκαπούρη είχαμε 20. Στον τομέα των επενδύσεων φαίνεται σαφώς στους διαπραγματευτές ότι η προσπάθεια είναι να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές όχι μόνο στην πρακτική των κρατών μελών, αλλά και στην πρακτική άλλων μεγάλων εμπορικών μας εταίρων. Και οι ε, ε, εταίροι μας μπορεί να επιμένουν στο ISDS με τις άλλες χώρες. Κάθε φορά που πείθουμε μια χώρα να δεχτεί το ICS τους κερδίζομαι και σε μία ε, μεγαλύτερη μάχη, δηλαδή να, ε, να ισχύει το ISDS ε, και να εφαρμόζεται από περισσότερες χώρες. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε για τον κώδικα των πολυμερών επενδύσεων. Τώρα το Βιετνάμ συνεργάζεται. Μετά την έγκριση και την κύρωση της συμφωνίας ΣΕΣ, στο βαθμό που θα υπάρξει και η συνένεσή σας, θα ασκήσουμε πιέσει στο Βιετνάμ για να εργοποιηθεί περισσότερο. Τώρα, θα είμαστε βέβαιοι ότι σε πέντε χρόνια θα υπάρχει η σε αυτή η συμφωνία. Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα κάνουμε το παν από την πλευρά μας για να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Τώρα η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ε, ασχολείται πολύ εντατικά με αυτό το θέμα. Κάνουμε συζητήσεις, αλλά θέλουμε και εταίρους στο εγχείρημα αυτό. Και οι καλύτεροι εταίροι είναι εκείνοι που έχουν συμφωνίες ICS. Γι' αυτό ο Καναδάς είναι εξαιρετικός εταίρος, γι' αυτό η Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ θα γίνουν ε, επίσης ε, σημαντικές. Ε, και εσείς θα βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Θα έχουμε λοιπόν το Διεθνές Σύστημα ICS, αλλά διμερώς υπάρχει το παλιό ICS. Είναι μια πρόκληση να αλλάξει αυτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Ίσως να σας ενδιέφερε ότι περίπου πριν από ένα χρόνο Στην Ομοσπονδιακή, Γερμανία, ε, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υποβλήθηκε έτσι ασύλο από έναν μεγάλο επιχειρηματία του Βιετνάμ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε υπεξαιρέσει 13 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια στη χώρα του. Ε, οι μυστικές υπηρεσίες του Βιετνάμ όμως είχαν στοιχεία για την υπόθεση και τον ανείχνευσαν μπόρεσαν να τον φέρουν στο Βιετνάμ όπου ε, δικάστηκε αφού του η μήνυση και μπήκε φυλακή. Είναι σημαντική λοιπόν η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τη βεβαιότητα ότι υπάρχει και κάποια αξιοπιστία αλλά και εμπιστοσύνη από την πλευρά των εταίρων μας. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τους επενδυτές που ε, τηρούν την ε, εσωτερική, την εγχώρια νομοθεσία του Βιετνάμ. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να είμαστε απολύτως ε, αυστηροί και συνεπείς με τις αρχές αυτές και να σεβόμαστε και την τοπική νομοθεσία όπως και την τοπική παράδοση στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Σωστά, σωστά. Για την πρώτη υπόθεση, να είστε βέβαιος ότι το ανέφερε επανειλημμένο στο Βερολίνο αυτού το είδους τον εκβιασμό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά αμφίδρομα. σε όλη την γεωγραφική ζώνη της Κεντρικής Ασίας και της Νοτιοανατολικής. Θέλετε κύριε αντικαταστάτη του σκιώδους εισηγητή να πείτε κάτι. Ωραία. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και με τα σημεία 6 και 7. Και για τα δύο ε, τμήματα, το εμπορικό και το επενδυτικό. Θα πάει η αντιπροσωπεία μας στο Βιετνάμ 29 έως 31 Οκτωβρίου. Μετά θα επιστρέψουμε και στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα έχουμε επιπλέον ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας. Και μετά θα ορίσουμε και προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες στις 2 και 3 Δεκεμβρίου. Και την πρώτη, στην πρώτη συνεδρία του Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε και το Φεβρουάριο θα περάσει στην Ολομέλεια. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τώρα με το τμήμα της δημόσιας συνεδριασής μας. Και σε δύο ακριβώς λεπτά θα έχουμε τη συνεδρίαση των ε, συντονιστών σε μετακύληση.